con la necesidad de presentar las enmiendas con tiempo suficiente para que el ponente pueda hacer un paquete πρέπει να είναι μία οδηγία που δεν θα είναι μόνο η οδηγία της ενιαίας ε, άδεια. Θέλουμε να είναι πλήρες περιεχομένου. Πιστεύουμε ότι το κείμενο της Επιτροπής είναι βελτιώσιμο και πρέπει να βελτιωθεί. Η Επιτροπή Επασχόλησης ασχολήθηκε με τέσσερα κύρια θέματα που την απασχολούν. Έχουμε ε, 16 τροπολογίες καταθέσει. Τα τέσσερα θέματα που μας απασχολούν κυρίως είναι το εξή. Δεν είναι λογικό. Μια τέτοια οδηγία ίσης μεταχείρισης να αφήνει στα χέρια των κρατών μελών θέματα τόσο σημαντικό όσο είναι το θέμα τη προστασία. Βεβαίω, η κατάσταση της αγοράς κάθε κράτους μέλου είναι διαφορετική. Αλλά αν έχει σημασία αυτή η οδηγία είναι διότι δίδει κατά ελάχιστον κάποια δικαιώματα τα οποία πρέπει να είναι τα ίδια σε όλα τα κράτη-μέλη. Έχουμε πει το θέμα καταθέσει τέσσερι τροπολογίε. Η πρώτη αφορά του εργαζόμενου οι οποίοι μετακινούνται. Εάν ένα μετανάστης, εργαζόμενο πηγαίνει σε ένα κράτος μέλος να εργαστεί θα πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα τα εργασιακά με τα τα οποία έχει και οποιοδήποτε εργαζόμενος του κράτους υποδοχής. Το λέμε αυτό λοιπόν στην Επιτροπή και θα θέλαμε να το διευκρινίσει αυτό. Να λέει δηλαδή ότι στην οδηγία θα πρέπει τα θέματα αυτά να τα χειριστούμε με σαφήνεια ώστε να λέγεται ότι θα εγγυηθούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων οι οποίοι μετακινούνται από τη χώρα σε μια άλλη χώρα. Δεύτερο, η δεύτερη τροπολογία αφορά το 12.1β και πρόκειται για την τροπολογία μας 8 που αφορά θέματα φορολογικά. Εάν πληρώνουν την εφορία ε, στη χώρα στην οποία εργάζονται οι μετανάστες θα πρέπει να απολαμβάνουν των ίδιων δικαιωμάτων που απολαμβάνουν και οι πολίτες της χώρας αυτούς. Δεν ε, τίθεται θέμα αδικίας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Τρίτο θέμα. Επίσης ένα θέμα σημαντικό, τροπολογία 12 στο 12, όταν χάνει τη δουλειά του ένας μετανάστης, δεν ε, θα πρέπει ε, εκ, του, ε, εκ νέου να ξαναζητήσει να αποτελέσει μέρος συνδικάτου ή να μην έχει πλέον κανένα δικαίωμα ή το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Επίσης, τροπολογία 13. Όταν χάνει τη δουλειά του ένας ε, μετανάστης πρέπει να έχει όλα τα δικαιώματα τα οποία απολαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος. Τα επιδόματα ανεργίας, το, την ε, κοινωνική ασφάλιση, όλα τα δικαιώματα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία είχε όταν εργαζόταν. Αυτό στα πλαίσια της μεταχείρισης με τους ε, ίδιου πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είπε η κυρία Ματιό, για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την παράνομη ε, μετανάστευση, θα πρέπει να δίδουμε στους νόμιμους εργαζόμενους τα ίδια δικαιώματα που δίδουμε στους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικά δεν θα είμαστε συνεκτικοί στην πολιτική που θέλουμε να ακολουθήσουμε και θα καταστρατηγούμε τα δικαιώματα των ε, μεταναστών αυτών εργαζομένων. Σας ευχαριστώ κύριε Θέρκα. Θα ακούσουμε πρώτα απ' όλα την Προεδρία και μετά την Κομισιό, εάν θέλει να λάβει το λόγο. Η Ισπανική Προεδρία, παρακαλώ. Ο κύριος Δουένιας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Προεδρία δεν έχει να προσθέσει πολλά σε σχέση με την ε, τελευταία παρέμβαση που έγινε. Αυτό που είναι σημαντικό για το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή είναι να ξέρει ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου επί του παράγοντος κειμένου που εξετάζεται. Ξέρουν και οι δύο επιτροπές ποια είναι η θέση η οποία ε, έχει εγκριθεί από την πλειοψηφία των συναδέλφων μου στο Συμβούλιο. Επίσης θα ήθελα, έχοντας ακούσει την κυρία Ματιέ, ότι διαπιστώνουμε ότι η Επιτροπή σας έχει κατανοήσει πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό πόσο πολύπλοκο είναι. Απλώς θα ήθελα να επιμείνω στο εξής. Το θέμα της οδηγίας δεν είναι τόσο να δώσει στους αλλοδαπούς εργαζόμενους τα ίδια δικαιώματα με αυτά των οποίων χαίρουν οι κοινοτικοί πολίτες, αλλά όλοι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι να έχουν το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων, όποια και αν είναι η χώρα καταγωγής τους. Αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσω και να το έχετε κατά νου. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να πω βασικά ότι ότι το Συμβούλιο αναμένει την θέση του Κοινοβουλίου για να μπορέσει να αντιδράσει. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ η Κομισιό. Ε, euh, Καταρχήν, η Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει την κυρία Ματιέ για το σχέδιο εκθεσή τη, το οποίο είναι ιδιαίτερα ισορροπημένο και να την ευχαριστήσουμε επίση γιατί έχει τονίσει το γεγονό ότι τα επιπλέον έγγραφα που τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να προσθέσουν ως παράρτημα στην ενιαία άδεια θα πρέπει να έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό για την ισορροπία αυτής της πρότασης. Τώρα, όπως σωστά υπέδειξε η συγγήτρια, είναι μια πρόταση κλειδί για την οικοδόμηση που θέλουμε να είναι σταδιακή μια κοινή πολιτική για την μετανάστευση. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονό ότι βρισκόμαστε σε ένα χώρο πολύ ευαίσθητο και στο πλαίσιο αυτό έχουμε δύο προσδοκίε. Η πρώτη είναι να ξεκινήσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσει που έχουν μπλοκαριστεί εδώ και χρόνια, αυτό και επί τη βάση τη πρόταση τη Κομισιόν, λαμβάνοντα υπόψη φυσικά τι τροπολογίε του Κοινοβουλίου και επίση ορισμένε βελτιώσει στο κείμενα που είχαμε επιτάπητος πριν η Ισπανική Προεδρία να ασχοληθεί με το ζήτημα, κάποιες βελτιώσεις λοιπόν που θα ήταν αποδεκτές σε επίπεδο Συμβουλίου. Και μάλιστα, όπως υπογράμμισε η κυρία Ματιό, το πεδίο το ευρύ, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα για μας να φτάσουμε σε συμφωνία σε ευρύ πεδίο εφαρμογής που θα αφορά όχι μόνο τους ετούντες την ενιαία άδεια, αλλά όλους τους εργαζόμενους των χωρών που βρίσκονται στην Ένωση. Επίτα μεγάλη φιλοδοξία είναι να φτάσουμε σε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Πιστεύουμε πω είναι η κατάλληλη στιγμή για δύο λόγου. Καταρχήν, έχουμε μια νέα συνθήκη που στον τομέα αυτό μα επιτρέπει τη συναπόφαση και άρα επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να συμμετέχει πλήρως στην υιοθέτηση της πρότασης αυτής και να προσθέσει σίγουρα μια μεγάλη προστιθέμενη αξία. Δεύτερον, έχουμε μια πολιτική εντολή που μόλις υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, που είναι εξαιρετικά φιλόδοξο όσον αφορά την νόμιμη μετανάστευση. Έχουμε ως στόχο έχει οριστεί μάλλον ο στόχο να επεξεργαστούμε μέχρι το 2013-2014 ένα κώδικα μετανάστευση. Δηλαδή να παγιωθεί αυτό το σύνολο που φαίνεται να είναι ανομοιογενέ και άνισο αλλά προς αυτό ε, κατευθυνόμαστε. Και για να απαντήσω στην κυρία Ματιέ, η Κομισιόν έχει την πρόθεση να απαντήσει ε, με δύο προτάσεις πριν από το καλοκαίρι για τους εποχιακούς εργαζόμενους και για τους ε, εργαζόμενους που είναι αποσπασμένοι στο εσωτερικό ενός ομίλου εταιριών, ICT είναι η στα αγγλικά. Είναι προτάσεις οι οποίες αφορούν τους όρους εισδοχή, διευκολύνσει για αυτές τις δύο κατηγορίες εργαζομένων. Τώρα, ε, για να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, η πρόταση αυτή, η πρόταση για την ενιαία άδεια είναι μια βασική, ένας βασικό στάδιο για μας μέσα σε αυτήν την σταδιακή δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου όσον αφορά την μετανάστευση. Ε, ήδη συμπεριλαμβάνει διάφορες πρόοδους, δεν θα πρέπει αυτό να το παραβλέψουμε. Φυσικά η Κομισιόν είναι έτοιμη να ευνοήσει κάθε δυνατή συμβαστική λύση ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο ώστε να διασφαλίσει ότι αυτός ο στόχος στον οποίο οποίο έχουμε κενό με την εισηγήτρια, δηλαδή η οθέτηση στην πρώτη ανάγνωση να υλοποιηθεί. Σας ευχαριστώ. Merci. Tenemos ahora algunos eh, miembros. Κάποιοι συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Πρώτα απ' όλα η κυρία Μπίνκεβιτσιούτε. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Βερονίκ Ματιού για την έκθεση την οποία παρουσίασε και ελπίζω πραγματικά να ε, τύχει της συνένεσης της Επιτροπής Απασχόλησης και του Συμβουλίου έτσι ώστε στην πρώτη ακρόαση να καταλήξουμε σε συμφωνία. Το άρθρο 29 της Συνθήκης της Λισαβόνας ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, καθορίσει μια κοινή ε, ε, πολιτική απασχόλησης και ότι θα πρέπει να εδραιώσει ισότιμα δικαιώματα ή με δαπών και αλλοδαπών εργαζομένων στη χώρα αυτή, στη χώρα υποδοχής. Υποστηρίζω και συμφωνώ με την εισηγήτρια η, οποία πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο των ισότιμων ε, μέτρων θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την ελαφραία μετανάστευση και εργασία. Θα μπορέσουμε επίσης να απλοποιήσουμε τα διοικητικά μέτρα και την γραφειοκρατία. Είμαι και σκιώδης εισηγήτρια και θα ήθελα να, σας, να κάνω μερικές παρατηρήσεις το πιο σημαντικό είναι οι εποχιακά εργαζόμενοι και αν θα καλύπτονται ή όχι από το πεδίο ισχύω της οδηγίας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νομική βάση, νομικές πράξεις στην Ευρώπη οι οποίες να, ορίζουν το καθεστώς των εποχιακά εργαζομένων και την, το νομικό τους καθεστώς. Ακούσαμε πολλά να λέγονται από αυτού του θέματος. Μας υποσχέθηκαν ε, προτάσεις ε, επί του εγγράφου αυτού. Το ακούσαμε και από την Κομισιόν και συζητήσεις έχουν γίνει από το 2007 αλλά ακόμα δεν έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Το τρίτο τμήμα του εγγράφου που συζητούμε λέει για τα ισότιμα δικαιώματα και ότι ελάχιστα πρότυπα, ελάχιστα στάνταρτς θα πρέπει να ε, καθιερώνονται. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τους εποχιακά εργαζόμενους. Για όλους να ισχύει και για εκείνους που εργάζονται εποχιακά. Έχω να, θα ήθελα να ρωτήσω την εισηγήτρια για τους πρόσφυγες και τα δικά τους δικαιώματα όσον αφορά τη συμπερίληψή τους στο πεδίο ισχύω. Ίσως θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για την τροπολογία 28. Γιατί πιστεύετε ότι δεν θα πρέπει το πεδίο να καλύπτει τους ε, πρόσφυγες. Επίσης την τροπολογία 52 όσον αφορά την τροπολογία 52. Το άρθρο 29 της συνθήκης της Λισαβόνας λέει ε, αναφέρεται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές για την απασχόληση ε, ημεδαπών ε, κλπ. κλπ. Δεν κατανοώ ακριβώς το περιεχόμενο της τροπολογίας 52. Θα ήθελα μερικές ε, αποσαφηνήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπόσκουρτ. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω μία σύντομη ερώτηση. Γιατί η διασύνδεση της άδειας παραμονής ε, με την άδεια εργασίας είναι ακριβώς το ζητούμενο εδώ. Είναι, το, ε, είναι σαφής αυτή η διασύνδεση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την κυρία Ματιού. Ματιού. Ε, πώς, ε, αν θα καλυφθούν ή όχι οι, τα μέλη της οικογένειας ε, τα οποία ήρθαν ε, υπό το καθεστώς της επανένωσης των οικογενειών ε, για, τους προσκάλεσε ο αλλοδαπός εργαζόμενος σε μια χώρα και ήρθαν ως μέλη της οικογένειας του. Ε, τι θα γίνει με αυτά τα μέλη μιας οικογένειας που ήρθαν σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την ε, διευκόλυνση της επανένωσης οικογενειών. Εμπίπτουν στο πεδίο ισχύω ή όχι. Ο κύριος Ντεβέρ όχι ακόμα. Η οχι ο κυριος ντεβερα οχι Κίνγκα Καλ. Ευχαριστώ. Αφενός, συμφωνώ. Αφενός θα πρέπει να συμβενήσουμε όλοι ότι πρόκειται για ένα, μια πάρα πολύ σημαντική νομοθετική πράξη. Ίσως και μετά την πρώτη αναγνώση θα μπορούσαμε να καταλήξουμε συμφωνία. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή μας σε αυτό το οποίο μας είπε η Ισπανική Προεδρία. Δεν πρόκειται για την χορήγηση των ίδιων δικαιωμάτων στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλους τους αλλοδαπούς, αλλά να χορηγήσουμε τα ίδια δικαιώματα σε όλους τους αλλοδαπούς εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι σημαντικό, διότι δεν την χάνουν τις ίδιες μεταχείρισης οι εργαζόμενοι. Ούτε καν στην ε, ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ υπηκόων νέων και παλιών κρατών μελών, αν μπορώ να το πω έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως αυτό το οποίο είπε η Προεδρία. Επίσης, φαίνεται ότι υπάρχει, από ό,τι μας είπε και εκπρόσωπος του Συμβουλίου, κάποια συμφωνία μεταξύ κρατών μελών και Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε σύντομα να καταλήξουμε σε συμφωνία. Υπάρχει και το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Ε, προβλέπεται ε, μία τριετής προθεσμία και θα ήθελα να προτείνω να ακολουθήσουμε αυτά τα οποία λέει το Συμβούλιο. Η κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα αένα, πρόβλημα της ε, προφοράς των, των ονομάτων σωστά. Έχουμε και τις σκοτσέζικες ιδιαιτερότητες. Εν πάση περιπτώσει, λέει η κυρία Λάμπερτ, έχω ορισμένες παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά στους πρόσφυγες και σε αυτά τα άτομα αυτά που χρειάζονται και χαίρουν ενός καθεστώτος προστασίας, διεθνούς προστασίας. Τώρα θα πρέπει να ρωτήσω, μέσα σε ποιο πλαίσιο παροχής ε, δικαιωμάτων θεωρούμε τους πρόσφυγες, ότι εμπίπτουν οι πρόσφυγες. Εγώ πιστεύω ότι αν συζητούμε για άτομα τα οποία χαίρουν ενός καθεστώτος διεθνού προστασίας, τότε αυτά τα άτομα δεν θα πρέπει να καλύπτονται από το πεδίο ισχύω. Αλλά εάν συζητούμε για άτομα τα οποία ε, πρέπει να προστατεύονται και, που, οι, οποίοι, οι οποίοι εργάζονται διασυνοριακά, είναι, μπίπτω στο καθεστώς διασυνοριακών εργαζομένων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να εξετάσουμε. Και ε, αν πάλι ε, εξετάζουμε το πρόβλημα αυτό μέσα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας, τότε μπορούν να εμπίπτουν ε, στο πεδίο ισχύω. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια επιλογή και να διευκρινίσουμε ε, άτομα που εμπίπτουν σε ποιο καθεστώς καλύπτονται από το πεδίο ισχύω ε, και σε ποιους μπορούμε να, να δώσουμε ακριβώς, να παράσχουμε αυτή την ισότητα μεταχείρισης και την ενιαία άδεια. Πρέπει λοιπόν να, να διευκρινίσουμε ισότητα δικαιωμάτων, αλλά πάνω σε ποια βάση. Ε, δεν ε, λυπάμαι που προτείνεται η διαγραφή του εκτιμώντας 19 ε, εναντίον των διακρίσεων, διότι η καταπολέμηση των διακρίσεων αποτελεί θεμελιολήθο της, ε, του νομικού πλαισίου της, ε, νομοθεσί, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Πιστεύω ότι μπορεί το εκτιμώντας αυτό να ισχύει και για ε, τους εργαζόμενους, να καλύπτει άτομα που εργάζονται. Και γι' αυτό διαφωνώ με τη διαγραφή του. Επίσης, πρέπει να είμαστε σαφείς ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία στην πρόταση αυτή για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους. Κάπως έχω την εντύπωση ότι αυτή η πρόταση οδηγίας απλώς κωδικοποιεί προηγούμενες διατάξεις και να ε, υπάρχουν ήδη νομικό πλαίσιο. Πρέπει να ξέρουμε συγκεκριμένα ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτής της πρότασης οδηγίας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ήθελα τώρα να δώσω το λόγο πάλι στην κυρία εισηγήτρια κυρία Ματιό να απαντήσει στα σχόλια και στις παρατηρήσεις που έγιναν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ρώτησα λοιπόν την Κομισιόν για την συμπερίληψη όχι ενός ε, πεδίο εφαρμογή για του αποσπασμένου εργαζόμενου και του εποχιακού εργαζόμενου. Η απάντηση ήταν σαφή ότι θα έχουμε προτάσει πριν το καλοκαίρι και γι' αυτό το λόγο δεν του έχουμε συμπεριλάβει στην ε, έκθεση αυτή. Το ίδιο ισχύει και για τους πρόσφυγες. Δεν είναι, εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογή για τον απλούστατο λόγο, αλλά εδώ θα ξαναθέσω την ερώτηση στην Κομισιόν, Από όσο γνωρίζω θα υπάρξει ένα σχέδιο ε, πρόταση της Κομισιόν για τους πρόσφυγες. Γι' αυτό το λόγο δεν θεωρήσαμε πως έπρεπε να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογή αυτής της πρότασης οδηγίας. Τώρα, στο πεδίο εφαρμογή και για την οικογενειακή επανένωση. Θεωρούσα ήδη πως ήταν λογικό να αναφέρουμε τα άτομα αυτά στο πεδίο εφαρμογή γιατί είναι άνθρωποι που εργάζονται, δεν έχει σημασία αν εμπίπτουν στι ίδιες κατηγορίες ή όχι, δεν νομίζω πω στο Συμβούλιο δεν δημιουργήσε πρόβλημα, ούτε και σε εμά δημιουργεί πρόβλημα. Είναι άνθρωποι που εργάζονται και δεν έχει σημασία για ποιο λόγο έφτασαν ε, αρχικά οι άνθρωποι αυτοί στην Ευρώπη. Εκτό αν βέβαια για εσά είναι πρόβλημα. Εγώ δεν κατάλαβα καλά την Τζίνα. Δεν κατάλαβα ακριβώς το θέμα του εκτιμώντας εννέα. Μήπως μπορεί να μου το ξαναπεί. Αν υπάρχουν άλλε ερωτήσει, είμαι στη διάθεσή σα. Θέλετε να κάνετε κανένα συμπληρωματικό σχόλιο, κύριε Σέρκα. Όχι. απλώ θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δώσατε να σα εξηγήσω αυτό που ήθελα. απλώ και να ζητήσω στους συναδέλφους να εξετάστε θετικά τις προτάσεις μας και αν μπορέσουμε να έχουμε διάλογο μεταξύ ημών, ημών και του Συμβουλίου να τον κάνουμε συντονισμένο τρόπο. Εγώ άκουσα τι είπατε. Σε κάποια θέματα συμφωνώ περισσότερο από τις άλλα, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να κάνουμε και οι τρεις κάτι πολύ καλό συνεργαζόμενοι προς καλό όλων. Υπάρχει καμιά παρετέρω διευκρίνηση, κυρία Μπόσκουρτ. Ευχαριστώ. Μία συμπληρωματική ερώτηση που αφορά τα μέλη των οικογενειών. Κατά τη γνώμη σας, λοιπόν, πρόκειται μόνο για άτομα τα οποία εμπίπτουν στο πλαίσιο της επανένωσης των οικογενειών, οι οποίοι έρχονται ε, στη χώρα υποδοχής και θέλουν να εργαστούν. Ναι, αλλά αν πρόκειται για, μια, για ένα ηλικιωμένο άτομο, μια γιαγιά ας πούμε, η οποία δεν θέλει να εργαστεί, ούτε δεν μπορεί, ε, δεν πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Εγώ ε, δεν, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Κυρία Ματιού. Κοιτάξτε, η άδεια ενιαία είναι άδεια παραμονής και εργασίας. Δηλαδή από τη στιγμή που πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα που δεν εργάζεται, δεν θα έχει αυτή την ενιαία άδεια την μοναδική αυτή άδεια. Ε, δεν, μπορεί να, δεν μπορεί να κάνει αίτηση για άδεια εργασία. Περιμένουμε να ακούσουμε την Κομισιόν. Άρα δεν αλλάζει το στάτους του ανθρώπου. Μπορεί να μείνει, ακόμα και αν δεν εργάζεται. Thank um, Κομισιόν, ευχαριστώ, Πρόεδρε. θα πρέπει να δούμε την αρχική πρόταση της Κομισιόν που συμπλήρωσε η κυρία Ματιέ με πολύ καλό τρόπο. Το θέμα είναι ότι έχουμε διπλό πεδίο εφαρμογή στην πρόταση. Δηλαδή, έχουμε τους ανθρώπους που μπαίνουν στα κράτη-μέλη ε, που σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και που μπορούν να ακολουθήσουν αυτή την ενιαία διαδικασία και να πάρουν την ενιαία άδεια. Αυτό είναι για τους εργαζόμενους. Ανθρώπους που έρχονται για να δουλέψουν που χρειάζονται να δουλέψουν. Και έπειτα υπάρχει η άλλη διάταξη που περιλαμβάνεται στην πρόταση που λέει ότι αν ένα άνθρωπος, ε, επικόστη της χώρας, ε, έχει μπει είτε ως φοιτητή, είτε ως ε, μέλος της οικογένειας το οποιοδήποτε άλλο είδος ε, πλάνο υποδοχής στο κράτος μέλος και είτε σύμφωνα με εθνικούς κανόνες είτε σύμφωνα με το κεκτημένο της ε, Ένωσης έχει το δικαίωμα να εργαστεί τότε το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να αναγράφεται στην άδειά τους δεν αλλάζει το στάτους δηλαδή Απλώ τα κράτη-μέλη θα πρέπει να, το, αναγράφουν στην άδεια το αν επιτρέπεται ή όχι να εργαστεί το συγκεκριμένο άτομο και υπό ποιες συνθήκες. Για παράδειγμα, έχουμε έναν ε, μία σύζυγο που έρχεται να βρει το σύζυγό της που ήδη εργάζεται στην Ένωση, σύμφωνα με το κεκτημένο, είναι η... ο κανονισμός του 86 του Συμβουλίου θα της επιτραπεί να εργαστεί μετά από 12 μήνες. Δηλαδή μετά από 12 μήνες το κράτος μέλος θα γράψει στην άδεια τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται να εργαστεί το συγκεκριμένο άτομο. Δεν αλλάζει όμως το καθεστώς. Αυτό είναι για να, για το έχουμε προβλέψει για να είμαστε δίκαιοι προς το συγκεκριμένο άτομο, να γνωρίζουν ακριβώς πότε και μπορούν να εργαστούν και για τον επιθεωρητή εργασία ή έναν αστυνομικό που ελέγχει την ταυτότητα, την άδεια, να γνωρίζει αν αυτός ο άνθρωπος εργάζεται νόμιμα ή όχι. Αλλά σίγουρα δεν πρόκειται για αλλαγή καθεστώτος. Απλώς πρόκειται για αναγραφή των δικαιωμάτων που ήδη ισχύουν υπό την εθνική ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και ακόμα μια κουβέντα να πω για τους πρόσφυγες. Η Κομισιόν δεν θέλησε στην αρχική της πρόταση να συμπεριλάβει τους πρόσφυγες στο πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων. Όχι της ενιαίας άδεια, αλλά στο άρθρο περί δικαιωμάτων, δηλαδή το άρθρο 12 για το οποίο είναι υπεύθυνη η Επιτροπή Απασχόλησης. Για τον απλό λόγο ότι ήδη υπάρχει κεκτημένο κοινοτικό για τους πρόσφυγες. Είναι η πράξη 2004-83 για την... Πρόκειται για την οδηγία των προϋποθέσεων εκεί συμπεριλαμβάνονται διάφορα δικαιώματα των προσφύγων ε, και τα δικαιώματα αυτά θα έλεγα ότι είναι πιο ευνοϊκά από αυτά που προβλέπονται από αυτήν εδώ την πρόταση. Οπότε εμείς εδώ ως Κομισιόν θεωρήσαμε ότι τα δικαιώματα ενός πρόσφυγα που εργάζεται ήδη καλύπτονται από την κοινωτική νομοθεσία και θα δημιουργεί το σύγχυση ανάμεσα στα διάφορα μέσα, αν τους περιλαμβάνομαι και εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, νομίζω πως αρκούν αυτά. Ωραία, λοιπόν, ολοκληρώνουμε την εξέταση του σχεδίου έκθεση. Θα σα θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι στι 23 Μαρτίου το μεσημέρι στην Επιτροπή Λίμπη. Για την Επιτροπή Απασχόληση είναι 24 Μαρτίου. Αλλά όσον αφορά εμά, την Επιτροπή Λίμπη, Έχουμε ε, προθεσμία 23 Μαρτίου το μεσημέρι. Περνάμε τώρα στο σημείο 3. Άσυλο. Πολύ περίπλοκο θέμα. Έχουμε ένα σωρό πρωτοβουλίες εδώ και θα πρέπει να θυμίσουμε εξ αρχής πως έχουμε λίγο χρόνο και υπάρχει μια ολόκληρη δέσμη πρωτοβουλειών σε σχέση με το άσυλο εδώ. Καταρχήν έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Σημείο 4 όσον αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές και διαδικασίες στα κρατημέλη για τη χορήγηση αλλά και για την αφαίρεση διεθνού προστασία. Ένα ανανεωμένο κείμενο. Νέα διατύπωση. Προτείνω να ακούσουμε πρώτα την κυρία Γκυγιώμα που είναι η εισηγήτρια και μετά την Προεδρία και την Κομισιόν καθώς και θα ξεκινήσουμε και συζήτηση. Αλλά να σας θυμίσω παρακαλώ πως έχουμε τουλάχιστον πέντε πρωτοβουλίες εδώ σε σχέση με το άσυλο και ε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε χρονικούς περιορισμούς εξ αρχής. Κύριε Γκυγιόμ, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να κάνω γρήγορα. Δύο λόγια για να ξεκινήσω και να μιλήσω για το πλαίσιο εντό το οποίο εμπίπτει αυτή η πρόταση. Μεταρρύθμιση τη διαδικασία ε, για τις θεωρήσεις που ξεκίνησε σε μια ευρωπαϊκή φάση εναρμόνιση του ασύλου δεν ήταν επαρκή στο παρελθόν και άρα πολλοί συμφωνούν ότι πρέπει να γίνουν πολλές προσπάθειες. Επίσης θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, επανειλημμένες ε, επικρίσεις που ακούστηκαν για αυτό που από αποκαλείται ε, το λότο του δικαιώματος ασύλου και να ε, βελτιώσουμε την διατύπωση γιατί έτσι είχαμε διάφορα παραθυράκια που έδιναν ε, ευκαιρίες για διάφορες ερμηνείες εξαίρεσης. Σκοπεύουμε λοιπόν να καλύψουμε τα νομικά κενά και να συμβαδίσουμε και με την ε, νομολογία της ΣΕΝΤΕΑΣ. Ορισμένες τροπολογίες που θεωρούνται θεμελιώδης. στην ουσία κωδικοποιούν υποχρεώσεις οι οποίες ισχύουν μέσω του διεθνούς δικαίου και που μεταφράζονται και σε αποφάσεις στο δικαστηρίο όπως ας πούμε η ισότητα των μορφών αλλά και αποφάσεις που θα πρέπει να εκδίδονται μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσιο. Ευνοϊκά λοιπόν θα πρέπει να διακύμαθα καταρχήν στους ετούντες διεθνούς, διεθνή προστασία η εισαγωγή του δικαιώματος για την προσφυγή, για έσταση για δωρεάν δικαστική συνδρομή, η υποχρεωτική συνομιλία με τον ετών, ετούντα διεθνούς, διεθνή προστασία, αλλά και η προστασία των ιδιαίτερα ευάλωτων ετούντων. Εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι είναι λυπηρό που διατηρείται σε αυτό το κείμενο η έννοια της ε, ασφαλούς τρίτης χώρας με την εγκατάλειψη της ενιαίας, του ενιαίου ευρωπαϊκού καταλόγου και τη διατήρηση των καταλόγων των κρατών μελών. Κατά την άποψή μου αυτό δεν θα επιτρέψει να αποφύγουμε ορισμένες ανισότητες σε συνέπειες παρά την επεξεργασία στο κείμενο αυτό κριτηρίων και την τακτική επαλήθευση της κατάστασης ε, στις χώρες που θεωρούνται σίγουρες ή ασφαλείς. Οι δυσκολίες που μας περιμένουν απέναντι σε αυτό το κείμενο είναι Εξής. Καταρχήν πρόκειται για περίπλοκο κείμενο και η βάση ήδη το 2004 ήταν περίπλοκη. Στην πρώτη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών θα πρέπει να σου ομολογήσω πως η ιδέα μιας αναδιατύπωσης της αναδιατύπωσης ε, ε, προέκυψε ώστε να αλλάξει η ίδια η δομή του κειμένου. Η ιδέα ε, είναι βέβαια πολύ δύσκολη. Θα πρέπει ωστόσο να αναγνωρίσουμε πως αυτό το αρχικό κείμενο είναι αντικείμενο συμβιβασμού και υποχωρήσουν από τα κράτη-μέλη ώστε να υπάρξει ένα νέο σύστημα για τη χορήγηση ασύλου. Η δεύτερη δυσκολία είναι ότι πολλά κράτη-μέλη ε, δήλωσαν ότι είναι αντίθετα στις μεταρρυθμίσεις αυτές. Εν πάση περιπτώσει ότι έχουν δυσκολίες με κάποιες από αυτές τις μεταρρυθμίσεις που προτείνονται και κυρίως επειδή ε, αυτές θα σήμαιναν περισσότερο κόστος και διοικητικό φόρτο. Βέβαια οι οικονομικές επιτυχίες ε, είναι, έχουν μια λογική, αλλά εδώ μιλάμε και για αρχές και για ευθύνε των κρατών μελών. Με άλλα λόγια, αν ε, σκεφτούμε με την αγορά ασύλου, αν θέλουμε μάλλον να παραμείνουμε σε μια αγορά του ασύλου, καλύτερα να μην ασχοληθούμε με το θέμα. Έπειτα υπάρχει ένα πολιτικό παράδοξο, το αναφέρατε και εσείς πρόεδρε πριν από λίγο, ε, ότι πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο, ένα κείμενο το οποίο εντάσσεται μάλλον σε ένα γενικότερο, σε μια γενικότερη δέσμη. Πρόκειται για πέντε ε, προτάσεις οι οποίες είναι ε, στην ίδια δέσμη, όμως οι συζητήσεις δεν προχωρούν στον ίδιο βαθμό, με τον ίδιο ρυθμό στο Συμβούλιο και γι' αυτό είναι περίπλοκο αλλά και απαραίτητο να φτάσουμε σε μια συμφωνία οριζόντια για το σύνολο της δέσμης αυτής. Και ίσως η Κομισιόν και το Συμβούλιο μπορούσαν να μας διαφωτίσουν εδώ εγώ θα σταματήσω σε αυτά για την ώρα και ίσως να παρέμβω στο τέλος του γύρου της ε, τραπέζης και να σας δώσω ε, κάποιους προσανατολισμούς και το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούργος από πλευράς της Προεδρίας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε με ε, τον συγητή, με την εισηγήτρια ότι είναι ο θεμέλιος λίθος όλου του συστήματος διότι καταγράφει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι εγγυήσεις μπορούν να δοθούν στους ετούντες άσυλο. Πρόκειται για μία πάρα πολύ φιλόδοξη πρόταση και θα πρέπει να μελετήσουμε εμπεριστατωμένα το όλο θέμα στο Συμβούλιο. Άκουσα επίσης πώς αντιμετωπίζει το θέμα στο Κοινοβούλιο Συγγετρία. Πρέπει να σας πω ότι στο Συμβούλιο σε πολιτικό επίπεδο έγινε μια παρουσίαση, έγινε μια γενική ανταλλαγή απόψεων καταρχάς και είδαμε ότι υπάρχουν δύο αρχές που απορρέουν από την όλη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, οι υπουργοί θέλουν να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο εγγύσεων και δικαιωμάτων, έτσι όπως αντιστοιχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη, και συγχρόνως θέλουν η όλη διαδικασία να είναι αποδοτική, αποτελεσματική. Δηλαδή, θα μην γίνει επαχθής τόσο η γραφειοκρατία που να μας εμποδίσει από το να βρούμε μία γρήγορη λύση σε κάθε πρόβλημα. αλλά συγχρόνω, να μην είναι η όλη διαδικασία ελκυστική για αυτούς οι οποίοι θέλουν να την καταχραστούν. Αυτά συμπεράναμε μετά από την πρώτη συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο. Μετά άρχισαν οι συζητήσει σε τεχνικό επίπεδο. Και έχουν ήδη γίνει διάφορες συνεδριάσεις της σχετικής ομάδας που έλεγε το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Βεβαίως, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η θέση του Συμβουλίου και πιστεύω ότι θα καθυστερήσουμε κάποιο χρόνο. Δεν λέω μέχρι να, φτάσουμε και σε, μέχρι φτάσουμε και σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο. Πιστεύω όμως ότι πρόκειται για μια, ένα σημαντικό θέμα και θα πρέπει να έχουμε μια εμπεριστατωμένη άποψη όλοι για να μπορέσουμε και τα τρία όργανα να καταλήξουμε σε οριστική θέση. Και δεν είναι θέμα ε, το οποίο θα μπορέσει να επιληθεί μόνο κατά τη διάρκεια μίας εξαμηνιαίας ε, προεδρίας. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία ανέφερε και η συγγήτρια απαιτούν να μελετήσουμε το όλο θέμα πολύ πιο προσεκτικά και να συνεχίσουμε τις τεχνικές συζητήσεις πριν να διαμορφώσουμε θέση. Σφαιρικά όμως πρέπει να πω ότι είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε μαζί σας και να φτάσουμε σε συμφωνία, σε συνεννόηση μαζί σας. Το σέλος δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Σας ευχαριστώ. Εκπρόσωπος της Επιτροπής, παρακαλώ. Η κυρία Μαρτίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε μια μεγάλη αντιπροσωπεία και μας εξόρισαν στο μέσον της αίθουσας. Αλλάξαμε θέση. Καταρχά, ε, λοιπόν, ευχαριστώ την συγγύητα κυρία Γκυλιόμ. Είχαμε αρκετέ συναντήσει ε, μαζί τη για, για διαβουλεύσει, για να συζητήσουμε μαζί τη ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο για να ενισχύσουμε ε, το πλαίσιο τη προστασία και τη ασφάλεια και για να καταλήξουμε σε, ένα, σε μια ισότιμη βάση αντιμετώπισης των ατόμων αυτών. Όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι πάρα πολύ φιλόδοξο κείμενο αυτό και οι διαβουλεύσεις επί του φακέλου αυτού θα είναι δύσκολες. Από τις τρεις δυσκολίες που τόνισε η συγγήτρια, ε, παραδέχουμε ότι είναι περίπλοκο κείμενο, η κυρία Γκυγιόμ, επισήμανε τους λόγους για τους οποίους ακριβώς είναι δύσκολο το κείμενο. Υπάρχουν εγγενείς δυσκολίες τις οποίες κληρονομήσαμε από προηγούμενα κείμενα. Επίσης συζητήσαμε το, τις δυσκολίες αυτές ήδη σε διμερείς συζητήσεις με τους κοιόδης εισηγητές. Η Ετέθη το θέμα της προστιθέμενης αξίας για την αναδιατύπωση των κειμένων. Πιστεύουμε ότι στην τρέχουσα οδηγία υπάρχουν θετικά στοιχεία τα οποία θέλουμε να διατηρήσουμε, θέλουμε να τα διαφυλάξουμε ε, στο, στην πρόταση οδηγίας. Δεν θέλουμε να ξανανοίξουμε τη συζήτηση σε κάθε σημείο και σε κάθε λεπτομέρεια. Γι' αυτό αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τα θετικά στοιχεία και να αναδιατυπώσουμε ορισμένα άλλα σημεία του κειμένου, επειδή ακριβώς είναι τόσο δύσκολο τόσο δύσκολος ο φάκελος. Βεβαίως έχουμε ανοιχτή προσέγγιση. Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε οποιασδήποτε δυνατότητες απλούστευσης του κειμένου και διευκρίνησης. Ε, η δεύτερη δυσκολία που είναι η αρνητική στάση πολλών κρατών μελών για την αναθεώρηση αυτή Βεβαίω, πολλέ διαβουλεύσει ήταν δύσκολε. Ούτε στο πρώτο κείμενο δεν ήταν εύκολε οι διαβουλεύσει που κάναμε με τα κράτη-μέλη Πήρα από πέντε χρόνια, όταν πρώτα παρουσιάσαμε την πρόταση. Όμω, εγώ προσωπικά σημείωσα ότι υπάρχει ένα, μια θετική προσέγγιση τώρα με ορισμένα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι όλα τα παλαιότερα κράτη-μέλη ε, υποστηρίζουν την πρόταση της ε, ισοτιμίας της, ε, και δεν επιθυμούν να διατηρηθούν οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με, την, ε, με τις ανισότητες που υπάρχουν στο πεδίο του ασύλου. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου, πρέπει να εξαλείψουμε αυτές τις διαφορές. Η τρίτη δυσκολία, που είναι αυτή η προσέγγιση πακέτο, Υπάρχουν πολλές προτάσεις στο τραπέζι που συζητώνται παράλληλα. Ορισμένα θέματα προς συζήτηση είναι οριζόντια και πρέπει να τα προσεγγίσουμε ε, συνεκτικά. Εμείς στην Κομισιόν προσπαθήσαμε βεβαίως να είμαστε ε, συνεπείς και συνεκτικοί στην πρότασή μας και να ανταποκριθούμε στις συζητήσεις που έγιναν και γίνονται στο Συμβούλιο. Αλλά και οι μελλοντικέ προεδρίες έχουν δεσμευτεί σε κοινή αντιμετώπιση και κοινή προσέγγιση αυτών των θεμάτων. Από ό,τι έχω ακούσει, το Κοινοβούλιο επίσης, το Ευρωκοινοβούλιο, ε, θα μελετήσει αυτά τα οριζόντια θέματα για να εξασφαλίσει ακριβώς τη συνέπεια μεταξύ των παράλληλων ενεργειών. Η προσέγγιση αυτή έχει τύχει θετικής ε, υποδοχής ε, και οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν με, τα, ε, με τους διάφορους συγητές, τους συναρμόδιους και στις διάφορες πολιτικές ομάδες για να καταλήξουμε σε μια κοινή προσέγγιση η οποία θα ωφελήσει την συνέπεια και τη συνοχή όλου του συστήματος. Ευχαριστώ, ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Μπορούμε να συζητήσουμε τώρα το θέμα αυτό. Ε, αλλά παρακαλώ να είστε σύντομοι. Είναι πέντε πρωτοβουλίες στο τραπέζι. Πρώτα, ε, η πρώτη ομιλήτρια η Μόνικα Χόλμαϊρ. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα δεν είναι καινούριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και και σε αυτή την ε, θητεία του σώματος και υπό την πίεση της Στοχόλμης προφανώς θα ερχόταν προς Υπάρχουν στοιχεία στην πρόταση τα οποία δεν δημιουργούν προβλήματα, τα οποία μπορέσαμε να διευθετήσουμε όπως ε, παραδείγματος η Eurodac, το Γραφείο για τους Πρόσφυγες και άλλα. Όμως υπάρχουν και προτάσεις οδηγιών που κατά την άποψή μου θα πρέπει να καλυφθούν, θα έπρεπε να είχαν καλυφθεί σε μία συνεκτική πρόταση. Το ότι έχουμε τώρα τρεις οδηγίες, μία για τις συνθήκες υποδοχής, μία για τα ελάχιστα πρότυπα, τρεις ε, για τα προσόντα που θα πρέπει να έχει να ε, υπάρχουν, να έχουν τα άτομα αυτά. Είναι τρεις ξεχωριστές οδηγίες και όχι μία όπου θα έπρεπε όλα αυτά να είχαν ε, καλυφθεί. Ε, οι τρεις αυτές διαφορετικές είναι οδηγίες και οι προτάσεις οδηγιών είναι αντιφατικές, δεν, είναι, δεν έχουν συνοχή, δεν έχουν συνέπεια και θα πρέπει να καλυφθούν από άπειρες διευκρινήσεις και ορισμούς. Διότι χρησιμοποιούν ορισμού διαφορετικούς που αναφέρονται στις ίδιες ε, ομάδες ατόμων. Εάν λοιπόν στόχος μας είναι να καλύψουμε ίδιες ομάδες ατόμων πρέπει οι ορισμοί αυτών των ομάδων να είναι ενιαίοι και όχι να διαφοροποιούνται. Έχω λοιπόν την, έχω την εντύπωση ότι οι ορισμοί οι διαφορετικοί ορισμοί επιτρέπουν ουσιαστικά τη μεγάλη διεύρυνση των ομάδων, των πληθυσμιακών ομάδων που εμπίπτουν στην πρόταση οδηγίας. Ε, φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο που πρέπει να αποφασίσουμε να ψηφίσουμε για την πρώτη οδηγία χωρίς να ξέρουμε ακριβώς σε ποιες πληθυσμιακές ομάδες απευθύνεται και ποιες καλύπτει. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ασυνέπεια και η ασάφεια των ορισμών. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε το θέμα των ορισμών ώστε να μην είναι αμφιλεγόμενοι, να είναι ξεκάθαροι και σαφείς πριν υπησέλθουμε στις διάφορες λεπτομέρειες των προτάσεων. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο το οποίο βρίσκω απαράδεκτο, ότι η, επίτροπο, η εκπρόσωπος της Κομισιόν λέει ότι δεν πρόκειται για αναθεώρηση ή για αναδιάρθρωση Εμείς πιστεύουμε ότι όπου πρέπει να γίνει αναθεώρηση πρέπει να το κάνουμε. Είναι και αυτό αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου. Εμείς, ε, εγώ θα ήθελα αυτά τα τρία θέματα τα οποία απευθύνονται στην ίδια πληθυσμιακή ομάδα, στην ίδια ομάδα τόμων να είχαν συμπεριληφθεί σε ένα πακέτο ώστε να μην έχουμε να κάνουμε με τρία κείμενα όπου το ένα παραπέμπει στο άλλο και τα τρία είναι περίπλοκα και έτσι δημιουργείται ε, μια τριπλή σύγχυση. Γι' αυτό ευχαριστώ την εισηγήτρια που ήδη από τώρα προσπάθησε να δημιουργήσει ένα συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών εισηγητών και των διαφορετικών πολιτικών ομάδων για να επιτευχθεί επιτέλους μια συμφωνία. Και τέλος, δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που λέει η εισηγήτρια ότι η η, αρχή, η πρόταση οδηγίας διέπεται από θεμελιώδεις αρχές και ευθύνες. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο το, θεωρητικό επίπεδο, υπάρχει και το οικονομικό επίπεδο, το, το ρεαλιστικό. Πρέπει λοιπόν η πρόταση, οι οδηγίες και όλες αυτές οι προτάσεις να είναι εφαρμόσιμες και να τις εξετάσουμε και από δημοσιονομική άποψη. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ε, πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις οι οποίες θα μας απασχολήσουν έντονα για το πώς ε, θα καταλήξουμε με τις τρεις αυτές οδηγίες, δηλαδή τις δύο που απασχολούν εμάς. Ευχαριστώ η κυρία Ενής Μα τι έγινε με αυτό το κινητό. Πρέπει να σας πω ότι αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα εδώ. Έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πακέτο προτάσεων. Έχουμε να κάνουμε κάποιες διαχωρισμό μεταξύ κάποιων ειδικών διαδικασιών και των υπολείπων θεμάτων. Εάν εγώ τώρα επικεντρωθώ στις διάφορες ε, συνθήκες ε, που πρέπει να επικρατήσουν στα πλαίσια των διαδικασιών, δεν βρίσκω λογική. Θα μπορούσα να αποδεχθώ τις τρεις ε, προτάσεις, αλλά όπως ήδη έχουμε ζητήσει από την Επιτροπή και μας το έχει άτυπα επιβεβαιώσει, καλύτερα θα ήταν να υιοθετήσουμε μία προσέγγιση οριζόντια. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να έχουμε τους ορισμούς και τις βασικές αρχές που χρησιμοποιούνται σε όλες τις προτάσεις, να συμφωνήσουμε επί όλων αυτών στο Συμβούλιο μεταξύ μας και μετά μεταξύ ημών του Συμβουλίου και της Κομισιόν και μετά να προχωρήσουμε στις τρεις προτάσεις για να προχωρήσουμε πιο εύκολα. Κατά την άποψή μου αυτή πρέπει να είναι η διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε. Διαφορετικά ε, ερχόμαστε μία πρόταση στην άλλη και προσπαθούμε να κάνουμε τι, να επανεφέρουμε τον τροχό. Εάν μπορούσε λοιπόν η Επιτροπή πρώτα απ' όλα να δει οριζόντια ποια είναι η προσέγγιση που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε πιο εύκολα να συμφωνήσουμε και εσείς μεταξύ σας και εμείς στο Κοινοβούλιο και τριμερός. Αυτά ήθελα να πω, χωρίς να μπω περαιτέρω σε λεπτομέρειες για τις διάφορες προτάσεις. Βεβαίως υποστηρίζω την εισηγήτρια και όλοι θέλουμε να υπάρχουν περισσότερες εγγύησεις, πιο αποτελεσματικές διαδικασίες, περισσότερα δικαιώματα και να μπορέσουμε την γραφειοκρατία κατά κάποιο τρόπο να την αποφύγουμε. Αυτό είναι λογικό. Απ' την άλλη όμω θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Και θα ήθελα να μου επιβεβαιώσει αυτό το οποίο μας είπε η Κομισιόν τώρα, καθώς και να μου πείτε, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, πότε μπορούμε να περιμένουμε τις διάφορες προτάσεις. Ευχαριστώ κύριε Μπουσούτιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπε η κυρία Χένη αυτά τα οποία ήθελα να πω. Θα είμαι λοιπόν πάρα πολύ σύντομη. Υποστηρίζω πλήρω τη δική τη έκκληση που γίνεται. Η προσέγγιση μα για το όλο πακέτο αυτό να είναι οριζόντια και είμαι υπέρ και τη προσέγγιση τη κυρία Μόνικα Χολμάιερ που εκφράστηκε πριν εάν δεν εντοπίσουμε πραγματικά τα κοινά θέματα που υπάρχουν μεταξύ όλων αυτών των ε, φακέλων οριζόντια, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, κύριε Πρόεδρε, εξετάζοντας το καθένα χωριστά και κάθε πρώτος χωριστά. Θα έλεγα λοιπόν ότι κατά κάποιο τρόπο χάνουμε το χρόνο μας εδώ, συζητώντας τις λεπτομέρειες της κάθε πρότασης χωριστά, πριν να έχουμε μια γενική ε, συνεκτική άποψη του όλου θέματος για να δούμε πώς συνδέεται μια πρόταση με την άλλη. Υποστηρίζω λοιπόν πλήρως τις απόψεις που εξέφρασαν οι συνάδελφοι προηγουμένως και τώρα. Πρέπει η Επιτροπή να μας βοηθήσει όντως για να εντοπίσουμε την ε, οριζόντια αυτή προσέγγιση και μετά ως Επιτροπή να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συνενετικές λύσεις επί αυτής της οριζόντιας πρόταση γενικότερα και μετά να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Okay, thank you. No more floors. Ευχαριστώ πολύ. Κανείς άλλος δεν θέλει το λόγο. Then, uh, yes, yes. Yes, please. Παρακαλώ. Madame Flotre. Ah, Κυρία Φλότχο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Σιλβή για με την παρουσία της και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει το όλο σκεπτικό για την πρόταση αυτή αναδιατύπωση της οδηγίας, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ σαφής και βασίζεται στην βούληση να βελτιώσουμε την όλη διαδικασία που αφορά το καθεστώς του πρόσφυγα. Θα πρέπει Συμφωνώ. Οι διαδικασίες να είναι πιο δίκαιες, πιο απλές για να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των προσφύρων. Μα λέει όμως το πρόεδρο του Συμβουλίου ότι αυτό είναι στόχος των Υπουργών. Εγώ βλέπω ποιε είναι οι επικρίσει που έγιναν στις συζητήσεις που έγιναν για αυτές τις προτάσεις στο Συμβούλιο Υπουργών τη 20 Νοεμβρίου και μπορώ να σα πω ότι για να μπορέσουμε στις δηλώσεις των κυρίων Υπουργών να διακρίνουμε μια κάποια βούληση να βελτιωθούν οι κανόνες με, για, που ισχύουν για τους πρόσφυγες μέσα των διαδικαστιών θα πρέπει πραγματικά να πάμε στην καφετζού, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Πιστεύω ότι όλο γραφειοκρατικές επικρίσεις ήταν προτάσεις. Λέουν ότι πρώτα θέλετε να, περάσουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των προσφύγων και μετά των πολιτών μας. Έγιναν λοιπόν πάρα πολύ έντονα σχόλια και δεν μπορώ να βρω καμία βούληση βελτίωση τη όλη κατάσταση. Και η κατάσταση όντω θα πρέπει να βελτιωθεί, κυρίω όσον αφορά τα κύρια σημεία τα οποία ανέφερε η συγγήτρια, η κυρία Σιλβιγκή που αφορούν ε, κάποια θέματα. Η το θέμα της ε, ε ανάκλησης ε, κάποιων ε, προσφυγών είναι πολύ σημαντικά, προσφυγή κατά κάποιες διαδικασίες δικαστική συνδρομή, όλα αυτά είναι θέματα πρωταρχικής σημασίας. Και πιστεύω ότι ούτως ή άλλως η πρόταση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πραγματικά έχει ως στόχο να βελτιώσει την κατάσταση των ατόμων που ζητούν προστασία. Τώρα, τα προβλήματα τα οποία ανέφερα Φερ, ε, η κυρία Κιγιώμ, ότι πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία. Το γεγονό ότι όλα αυτά είναι θέμα ενό πακέτου και ότι όλα αυτά είναι θέματα στη στο Συμβούλιο, είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα σκεφτούμε πάρα πολύ συγκεκριμένα. Βεβαίω, στι διάφορε προτάσει λέγω ότι θα πρέπει να βρούμε μια συνεκτικότητα. Υπάρχουν κάποιε έννοιε οι οποίε είναι κοινέ για όλε τι οδηγίε και θα πρέπει να τι ορίσουμε με ακρίβεια. Διερωτώ όμω, είναι η κατάλληλη στιγμή να διαφοροποιήσουμε τις διάφορες διαδικασίες, αν θα πρέπει να ασχοληθούμε πρώτα με όλες τις διαδικασίες ή θα πρέπει συγχρόνως να κάνουμε συζήτηση επί της ουσίας για την αναδιατύπωση ε, της οδηγίας εγκαρσίως διότι αν κάνουμε τα πράγματα πολύ τμηματικά, ίσως δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ε, συμφωνία για όλα αυτά τα κείμενα. Αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα που θέτω για θέματα αποτελεσματικότητα μιλώ. Αν ο στόχος μας είναι κοινό, θα βρούμε τρόπο να προχωρήσουμε με του καλύτερε δυνατέ συνθήκε. Δεν ε, με απασχολεί αυτό το θέμα τόσο. Θεωρώ ότι σήμερα ούτως ή άλλως θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τα κείμενα και να οργανώσουμε και εδώ θέλουμε μία πρόταση οργάνωση τη δουλειά, την οποία πρέπει να κάνουμε ώστε όσο προχωρούμε η συζήτηση των κειμένων αυτών και προχωρούμε στη συζήτηση στις διάφορες ομάδες και μεταξύ των σκιωδών εισηγητών να οργανωνόμαστε ώστε να κάνουμε συζητήσεις ε, προχωρώντας με τον ίδιο ρυθμό και κάνοντας τη δουλειά μας συνεκτικά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η οριζόντια ανάγκη συντονισμού ε, είναι σαφής. Ε, αυτό το είπαν πάρα πολλά μέλη ε, και συμμετέχονται στη συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια συζήτηση στο γυλής τραπέζης με το δίκτυο Οδυσσέους. Οδυσσέας και αυτό θα γίνει στις 26 Απριλίου 26 Απριλίου. Παρακαλώ σημειώστε το στεμερολόγιο ημερολόγιο σας τη συζήτηση αυτή των Αγγυλής Τραπέζης στις 1 η ώρα. 1 η ώρα το απόγευμα, 1 με 6.30. Α, όχι, 1 με 3 διορθώνει ο πρόεδρος. 1 με 3 το απόγευμα για να συζητήσουμε τα οριζόντια θέματα. Ας επανέλθουμε τώρα στην Επιτροπή και τη δίνουμε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Όλοι συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει συνέπεια και συνοχή. Δεν θα έλεγα όπως ε, είπε η κυρία Χολμάιερ ότι ε, θα πρέπει τις τρεις αυτές προτάσεις να τις αναδιαρθρώσουμε και να τις ενοποιήσουμε σε μία πρόταση. Θα ήθελα να θυμίσω ότι βάσει των διαθεσμικών συμφωνιών υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κανονισμοί. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα οριζόντιας φύσης, ναι, σύμφωνοι. Εδώ όλοι θέλουμε να διορθώσουμε τα στραβά. Αλλά δεν είναι μόνο οριζόντια τα θέματα οριζόντιας ε, διαχείρισης, αλλά οι τρεις προτάσεις αυτές είναι και πάρα πολύ διαφορετικές. Βεβαίως αποτελούν ε, τμήμα ενός πακέτου, αλλά έχουν διαφορετικούς στόχους. Ορισμένες φορές ε, οι ορισμοί είναι διαφορετικοί γιατί δεν ε, ε, καλύπτουμε αναγκαστικά ακριβώς τα ίδια άτομα. Ε, άλλοτε είναι πρόσφυγες, άλλοτε είναι ετούντες άσυλο. Γι' αυτό λοιπόν οι ορισμοί βρίσκονται εκεί που βρίσκονται και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εγώ δεν προσπαθώ να δικαιολογηθώ, θέλω να βοηθήσω. Θα πρότεινα λοιπόν οι εργασίες αυτές να γίνουν παράλληλα, δηλαδή οριζόντια προσέγγιση για λίγες, ε, λίγα θέματα, περιορισμένα θέματα, ας πούμε ορισμός οικογενειών, ε, διαδικασία αιτήσεων ε, κλπ. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα τα οποία πρέπει να συνεχιστεί η επεξεργασία τους, τα οποία δεν είναι οριζόντιας φύσης. Γι' αυτό λοιπόν εκτός από την οριζόντια ε, επεξεργασία θεμάτων ε, πρέπει να συνεχίσουμε και την ε, ανάπτυξη των άλλων θεμάτων που περιλαμβάνουν στις τρεις προτάσεις. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος η κυρία Γκυγιόμ. Σύντομα γιατί Βεβαίω υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά υπάρχει και η συζήτηση που θα είναι πολύ σημαντική για την, το μέλλον αυτού του θέματος και του κειμένου. Εγώ συμμερίζομαι την ιδέα της αναζήτησης μια συμφωνίας με το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Δεν θα είναι και πολύ απλό βέβαια, αλλά πιστεύω πως θα πρέπει να το, να το προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Ταυτόχρονα εμείς στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξουμε πλήρως το ρόλο μας στον ε, διαθεσμικό διάλογο και να κάνουμε και αυτή τη δουλειά για τη διερεύνηση, την αναζήτηση συνένεση όσο γίνεται ευρύτερη εντό του σώματος. μια δεύτερη σειρά παρατηρήσεων. Θα μου επιτρέψετε να προσπαθήσω ε, να συνεχίσω παρόλα αυτά με τους σκεώδεις και με όσους θα θελήσουν να εργαστούν πάνω στα θέματα αυτά ε, και να εργαστούμε ε, για την καρδιά του και τον πυρήνα του κειμένου για να προσπαθήσουμε να ε, νοήσουμε το περίπλοκο αυτό κείμενο, αν και καταλαβαίνω τις παρατηρήσεις σας και έγιναν παρατηρήσεις και σε προηγούμενες συναντήσεις όσον αφορά την οριζόντια δομή όπως εξάλλου υπόθηκε και σήμερα. Αυτό το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Δεν έχω ιδέα για κάποια ιδέα για το πώς θα υλοποιηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα για, με βάση αυτά τα οριζόντια στοιχεία. Η Κομισιόν ίσως θα πρέπει αυτό να μας το πει. Πιστεύω ωστόσο ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να ορίσουμε αυτή τη συμφωνία με τους διάφορους συντονιστές, τους συζητητές και τους σκιώδεις ε, όσον αφορά τα οριζόντια θέματα. Το έλεγα ότι είμαστε στην αρχή μιας μακράς και περίπλοκης εργασίας και θα ήθελα να βασιστώ στην προσήλωση όλων για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα σας ευχαριστώ που μιλήσατε για την ακρόαση και το στρογγυλό τραπέζι, τραπέζι της 26 η Απριλίου αν και δεν ξέρουμε ακριβώς ακόμα την ώρα για να δουλέψουμε ακριβώς για αυτά τα οριζόντια ζητήματα που αφορούν το άσυλο. Νομίζω πως είναι μια πολύ σημαντική ε, συνάντηση που θα μας επιτρέψει να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα και ε, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, αυτή η επιφύλαξη για την οριζόντια προσέγγιση και η απάντηση της Κομισιόν που είναι ακόμα εκρεμής, αν πρέπει να κάνουμε μια προσέγγιση για το χρονοδιάγραμμα, εγώ είχα φανταστεί ότι θα γινόταν πιο γρήγορα τα πράγματα. Πάντως τελικά βλέπω πως πριν από το Σεπτέμβριο δύσκολα θα μπορούσαμε να έχουμε ε, κάποια έκθεση ενώπιον της Επιτροπής. Ε, εν τω μεταξύ όμως σας δουλέψουμε. Σας ευχαριστώ. Προχωράμε λοιπόν. Συμφωνείτε, προχωρούμε και πάμε στο σημείο 5. Ελάχιστες απαιτήσει για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκών τρίτων χερών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας και το περιεχόμενο της παρεχόμενης ε, προστασίας. Ένα διατύπωση, εκδοχή. Ε, νέα εκδοχή δηλαδή. Έχουμε μια πρόταση που στόχο έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της ε, σύνταξης νομοθεσίας περί ώστε να διασφαλιστεί ψηλότερη και πιο εναρμονισμένη ε, προστασία και προδιαγραφές αυτής. Προχωρώντας προς μια ενιαία Ε, έχουμε διάφορες τροπολογίες, όχι μάλλον όχι, τροπολογίες περιμένουμε να έχουμε, αλλά εδώ έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Και να σας θυμίσω Και το σχέδιο έκθεσης θα παρουσιαστεί στην συνεδρίαση της Λίμπιας στις 23 και 24 Ιουνίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψε. Θα ακούσουμε πρώτα την εισηγήτρια, την κυρία Τζιν Λάμπερτ. Συγγνώμη που πριν σας μπέρδεψα με τον Ζαν Λαμπέρ που δεν είναι ανύπαρκτος. Έχετε το λόγο. Εντάξει, ευχαριστώ. Um, okay, the, as has been... Όπως ελέγχθη, αυτό που μας απασχολεί εδώ είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε εμείς προστασία. And at that point, Parliament was consulted. Um, we are now... Ναι, ελάχιστες απαιτήσεις. Οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσεις. Qualification uh, requirements. Η οδηγία αυτή ως έχει καλύπτει τις απαιτήσει για το καθεστώς του πρόσφυγα απαιτήσει που πρέπει να ισχύουν και για παράπλευρη προστασία. Ε, δηλαδή συμπληρωματική προστασία για τα άτομα αυτά τα οποία δεν εμπίπτουν στο καθεστώς του πρόσφυγα βάσει του ΑΚ 51 της Γενέβης αλλά που εν πάση περιπτώσει δικαιούνται συμπληρωματικής προστασίας παραδείγματος είναι κοινωνικές ομάδες ε, τις οποίες αναφέρει η Σύμβαση της Γενέβης του 51 ε, και ένα άλλο στοιχείο το οποίο ε, καλύπτεται από την ισχύουσα οδηγία είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να όχι μόνο να είναι να έχουν την ηθαγένεια μιας χώρας αλλά μπορεί να είναι και απάτριδες ή άλλος ανηθαγενής άνευ δηλαδή ηθαγένειας και το ερώτημα που μας απασχολεί τι είδου προστασίας μπορούμε να παράσχουμε το Ευρωκοινοβούλιο είχε ορισμένες δυσκολίες με την παρούσα οδηγία τουλάχιστον με τη μορφή ως έχει και ε, γι' αυτό ε, προτείνουμε ακριβώς ε, την οδηγία αυτή για τις ελάχιστες απαιτήσεις οι οποίες θα καλύπτουν το κοινωνικό δίκτυο προστασίας της υπηρεσίας υγείας αυτών των ατόμων. Παναδιατύπωση λοιπόν, αναδιάρθρωση της οδηγίας αυτής χρειάζεται διότι έχουν αλλάξει ορισμένοι ορισμοί. Και αυτή η αναδιατύπωση είναι αναγκαία γιατί υπό το πλαίσιο της αναθεώρησης διαπιστώσαμε ότι το καθεστώς αυτό προστασίας δεν είναι ε, αναγκαστικά ε, βραχυχρόνιο. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες, έχουν αλλάξει οι καταστάσεις βάσει νεότερης νομολογίας και γι' αυτό χρειάζεται ακριβώς αναδιατύπωση ορισμένων σημείων, ορισμένων προβληματικών διατάξεων ε, της ε, παλαιότερης οδηγίας. Κατά την άποψή μου, αυτή η πρόταση η οποία υπάρχει μπροστά μας είναι γενικά θετική, ε, παρόλο που δεν πηγαίνει όσο μακριά θα ήθελα εγώ. Δεν, δεν είναι τόσο δηλαδή ε, αποτελεσματική όσο θα επισημούσα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τα άτομα αυτός δικαιούχους διεθνούς ε, προστασίας παρόλο που υπάρχει και η κατηγορία του πρόσφυγα βεβαίως και να προσπαθήσουμε να ε, εναρμονίσουμε το καθεστώς προστασίας ε, ε, για αυτές τις ε, δύο κατηγορίες και ώστε να μην υπάρχουν αντιφάσεις και να μην σημειώνονται κενά στην παροχή προστασίας των ατόμων αυτών. Επίσης δεν θα πρέπει να δυσκολεύεται η πρόσβασή του στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στην αγορά εργασίας γι' αυτό πιστεύω ότι η πρόταση σε αυτό το σημείο περιλαμβάνει πάρα πολλά θετικά σημεία. Επίσης, αναφέρεται σε θέματα ορισμού ορολογίας, όπως παρατήρησαν και άλλα μέλη προηγουμένως, για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών που ενδεχομένως να χρειάζονται προστασία υπό το, την, το πλαίσιο της διευρυμένης οικογενειακής προστασίας ε, ιδίως για ε, άτομα τα οποία είναι ανήπαντρα ε, και επίσης χρειάζονται ορισμένες αναδιατυπώσεις σε άτομα τα οποία υπόκεινται διακρίσεις ή διώκονται λόγω του φίλου τους ή όπου επισέχεται το θέμα τη διάστασης του φιλου also... Και επίσης η αναδιατύπωση αυτή προσπαθεί να διευκρινίσει τον καλύτερο ορισμό της παρεχόμενης προστασίας στη χώρα η οποία την παρέχει, δηλαδή αποτελεσματική προστασία. Πώς είναι, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να υλοποιηθεί αυτό το πλαίσιο προστασίας. Ε, μην ξεχνάμε ότι υπήρχε ένα δίκτυο προστασίας ε, διεθνών δυνάμεων, ας πούμε στη Στρεμπενίτσα, το οποίο κατέρευσε και απέτυχε παταγωδός. Άρα λοιπόν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αποτελεσματική εφαρμογή της προστασίας αυτής. Υλοποίηση, σωστή υλοποίηση. Αυτή η αναδιατύπωση λοιπόν πιστεύω ότι θα είναι αναγκαία. Ακούσαμε πολλές παρατηρήσεις και διάφορες, διαφορετικές απόψεις. Γι' αυτό καλό θα είναι να διοργανώσουμε μία συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητής, δεδομένου ε, ότι υπάρχουν παράλληλες ε, οδηγίες εδώ που συζητιούνται και αυτά είχα να πω προς το παρόν ως εισαγωγικές παρατηρήσεις. Ε, Ευχαριστώ κύριε Λάμπερτ. Ισπανική Προεδρία παρακαλώ. Πάλι ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μας φαίνεται ότι είναι κλειδί αυτή η οδηγία για την όλη διαδικασία συλλού. Είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Από τεχνική πλευρά είναι λιγότερο πολύπλοκη, αλλά πρόκειται για ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλο το σύστημα ασύλου που θέλουμε να συστήσουμε. Η παρούσα οδηγία εγκρίθηκε κάτω ομοφωνία και μετά πρέπει να σου πω ότι έγιναν επί αυτού τις συζητήσεις επί του Συμβουλίου. Τώρα είμαστε στη διαδικασία της συναπόφασης και πιστεύουμε ότι όντως τα τρία θεσμικά όργανα μπορούν να κατρέξουν συμφωνία. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, όπως και για την προηγούμενη, αλλά με ένδειξη καλή βούληση εκ μέρους τόντων, αναμφίβολα θα φτάσουμε σε συμφωνία. Τώρα, η κατάσταση αναφορά τη διαδικασία είναι παρεμφερείς με αυτή που περιέγραψα στην προηγούμενη, για την προηγούμενη. Ήδη έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση, μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών και τώρα γίνονται τεχνικού επίπεδου συζητήσεις. Έγιναν διάφορες συναντήσεις, έχει γίνει ανάγνωση του κειμένου, υπάρχουν προβλήματα στα οποία θα πρέπει να εμβαθύνουμε για να τα ξεπεράσουμε. Ήδη υπάρχει μια αυτή η οδηγία εφαρμόζεται στα κρατημέλη και γι' αυτό όλοι με μεγάλη προσοχή βλέπουν οποιαδήποτε νέο μέτρο. Τώρα, θέματα που αφορούν ε, την ε, χώρα καταγωγής ή άλλα τέτοια θέματα, το επίπεδο της προστασίας, είναι θέματα τα οποία σχετίζονται καμιά φορά και με το κόστος και πολλές φορές έχουν σχέση με την τελική απόφαση που θα ληφθεί. Τώρα, τη χορήγηση του καθεστώτος ε, η αναγνώριση του δικαιώματος κάποιων υπηκών να ζητήσουν είναι επίσης θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και ακόμη δεν βλέπω να υπάρχει για αύριο η λύση. Φαντάζομαι όμως ότι θα, συνεχίσουμε ε, και μεταξύ μας μπορέσουμε ως θεσμικά όργανα και να συνεννοηθούμε, θα καταλήξουμε σε λύση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μιριέλ Γκάν, εκ μέρου του σε Επιτροπή. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τζιν Λάμπερτ για την ε, σφαιρικά θετική αξιολόγηση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπως είπε προηγουμένως και η Άντζελα Μαρτίνη, η αναδιατύπωση βασίζεται στην πρώτη εκδοχή της οδηγίας του 2004, δεδομένου ότι υπήρχαν στοιχεία θετικά, τα οποία συμπεριλάμβανε αυτή η οδηγία. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν κάποιες αδυναμίες όσον αφορά κάποιες, ε, κάποια ε, νομικά θέματα για θέματα νομικής ε, προστασίας στα πλαίσια της Σύμβασης ή σε πλαίσια άλλων συμβάσεων και χρειάστηκε να, να τα βελτιώσουμε. Επίσης, βασιστήκαμε στο πρόγραμμα της ε, στην ε, Σύμβαση του Ανθρώπινου Δικαιώματος, ώστε να δώσουμε ένα ενιαίο καθεστώς και να μπορέσουμε να έχουμε ενιαία ε, επίπεδο για τα δικαιώματα και την προστασία των δικαιούχων στα πλαίσια των ε, ελαχίστων απαιτήσεων επίσης πρέπει να πω ότι στις προτάσεις της η Κομισιό βοηθήθηκε από την εξέλιξη της κοινοτικής νομολογίας. Η Τζιν Λάμπερτ μίλησε για την πραγματική και μόνιμη προστασία. Εδώ και δύο εβδομάδες υπήρξε απόφαση του δικαστηρίου που επιβεβαίωσε κατά κάποιο τρόπο την πρόταση ε, της διατύπωσης στην οποία ακολούθησε για την αναδιατύπωση οδηγίας η Κομισιόν. Πρόκειται λοιπόν για ένα στοιχείο το οποίο μας ε, στήριξε και μας βοηθά να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά την προσέγγιση του καθεστώτος και την βελτίωση το περιεχομένου των δικαιωμάτων, εάν η συζήτηση δεν είναι τόσο ευαίσθητη η πολύπλοκη όσο και οι συζητήσεις για το άσυλο, σίγουρα θα γίνει εκτενή συζήτηση και για το θέμα αυτό. Ακούσαμε για κάποιες απόψεις κρατών μελών όσον αφορά το κόστος, όσον αφορά το κόστος για κάποια μέτρα που προτείνουμε. Τα συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα, τα αξιολογήσαμε στη μελέτη επιπτώσεων και πιστεύουμε ότι το κόστος αυτό είναι μικρότερο από ό,τι λέγεται σε κάποιες αναλύσεις. Θα ήθελα εξάλλου να υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο της Πρόσφυγης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, ταμείο αλληλεγγύης. Τελειώνοντας, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στις δύο προτάσεις ή στην οδηγία για την ε, διαδικασία ασύλου για τις ελάχιστες απαιτήσει δεν θα πρέπει να εξετάζονται κάθε μία μέσα σε στεγανά ή χωριστά δεδομένου ότι οι διάφορες εθνικές ε, διοικήσεις και η κοινωνία των πολιτών θα βοηθηθούν από το σχετικό Ευρωπαϊκό Γραφείο και θα μπορέσουν ε, να θέσουν τους πόρους τους από κοινού και να βελτιώσουν την όλη κατάσταση. Μπορούν λοιπόν σε συγκεκριμένη αυτή περίπτωση να γίνουν ακόμη και οικονομίες θα έλεγα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συζήτηση, κυρία Χολμάιερ, πρώτα απ' όλα. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Καταρχάς, μια σύντομη απάντηση στην ε, ανταπάντηση της εκπροσώπου της Κομισιόν. Κυρία Μαρτίνη, δεν ζήτησα τώρα μια νέα πρόταση η οποία αναδιέπεται από ε, συνοχή και συνέπεια. Ήθελα να την είχαμε αυτή ήδη στα χέρια μας. Όσον αφορά τώρα τις ε, απαραίτητες ε, προδιαγραφές ε, για την, την αναγνώριση, τις ελάχιστες επιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς, θέλω να, πω το, να ρωτήσω την Κομισιόν πότε θα είναι σε θέση να μας παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη αναδιατύπωση των ορισμών. Διότι είναι δύσκολο να προχωρήσουμε στις εργασίες μας εάν δεν έχουμε σαφείς ορισμούς στα χέρια μας. Πότε λοιπόν θα μπορέσει η Κομισιόν να μας παρουσιάσει τους σαφείς ορισμούς που είναι απαραίτητοι για να ξέρουμε ακριβώς ποια άτομα ποιου ορισμού εμπίπτουν σε ποιο πεδίο προστασίας δεδομένου ότι η νέα πρόταση οδηγίας προτείνει σημαντικές τροποποίησεις. Θα πρέπει λοιπόν όσον αφορά και τις διαδικασίες και τις δαπάνες να έχουμε σαφή ιδέα των ορισμών. Και προβλέπονται έντονες συζητήσεις. Άρα λοιπόν όλοι συμφωνούμε επί της αρχής ότι χρειαζόμαστε ένα ξεκάθαρο καθεστώς παροχής προστασίας το οποίο να καλύπτει άτομα τα οποία χρήζουν της προστασίας αυτής και να μην καλύπτει άτομα τα οποία δεν εμπίπτουν, δεν είναι κατάλληλα, δεν είναι επιλέξιμα και δεν χρειάζονται αυτή την προστασία. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν θα έχουμε συγκεκριμένους ορισμούς. Γι' αυτό έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και χαίρομαι για αυτές τις συζητήσεις που θα γίνουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Brown... Some people. Κύριος Μπρόνς, είπε ο πρόεδρος. Καλά. Ε, λοιπόν, όσοι, ε, όσοι ισχυρίζονται ότι είναι γνήσιοι ετούντες άσυλο, γλήσιοι ε, και σωστά ζητούν άσυλο, θα πρέπει να εξεταστούν βάσει των συγκεκριμένων ορισμών Ας μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι είναι ε, σωστοί, είναι πραγματικά άνθρωποι που ζητούν άσυλο και ότι είναι ειλικρινείς οι αιτήσει τους. Όμως ας μην ξεχνάμε επίσης ότι περνούν από διάφορες χώρες και ε, άρχισαν στην πρώτη χώρα υποδοχής την Οδύσσια τους ε, ως γνήσιοι ετούντες άσυλο, γνήσιοι πρόσφυγες αλλά η συνεχεία πηγαίνοντας από χώρα σε χώρα γίνανε οικονομικοί ε, μετανάστες ή οικονομικοί πρόσφυγες. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε και να υποδεχτούμε ολόκληρους πληθυσμού χωρών οι οποίες πλήγονται από πολέμους, από εμφύλιους πολέμους, από διαμάχες. Δεν μπορούμε να αγκαλιάσουμε και να δεχτούμε στις χώρες μας όλο τον πληθυσμό της υποσαχάριας Αφρικής ή ολόκληρες επαρχίες της Κίνας. Δεν λέω, υπάρχουν τυραννικά καθεστώτα όπου ε, εκατομμύρια ανθρώπων διώκονται και ταλαιπωρούνται και βασανίζονται. τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε, καταρχάς να σταματήσουμε να ταλαιπωρούμε δικούς μας πολίτες, Ευρωπαίους. Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σταματήσουμε να διεξάγουμε πολέμους εναντίον τρίτων χωρών. Ο πόλεμος κατά του Ιράκ παραδείγματος δημιούργησε πραγματικά ένα, μια χιονοστιβάδα από αυτούς τους ανθρώπους που εμπίπτουν στην κατηγορία των ετούντων άσυλο. Ευχαριστώ, κύριος Ντεγιόγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα σχόλιο θα ήθελα εγώ να κάνω, το οποίο αναφέρεται στις ε, παρατηρήσεις της Κομισιόν. Θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στο εξής. Πρέπει να αποφασίσουμε αν ζητούμε εδώ την καθιέρωση ενός πλαισίου προστασίας που θα έχει όρια. Θα έχει ορισμένα ανώτατα όρια, θα είναι οριοθετημένο. Δηλαδή μέχρι πού θα επεκτείνεται, μέχρι πού θα καλύπτει και θα παρέχει αυτή την προστασία. Αν δείτε το άρθρο 15, το οποίο ορίζει τι σημαίνει στα αγγλικά serious harm, σοβαρή βλάβη, σοβαρή ζημία. Ε, μπορεί ορισμένε άλλε χώρε να χρησιμοποιούν διαφορετικέ ερμηνείε και διαφορετικά κριτήρια, ιδίω όταν πρόκειται για συμπληρωματικά καθεστώτα προστασίας υπάρχει διακριτική ευχέρεια κρατών μελών να ε, χρησιμοποιήσουν διαφορετικούς ορισμούς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Αν θα είναι ενδεικτικό αυτό το πλαίσιο ή αν θα είναι ε, οριστικό, δηλαδή καταληκτικό. Από εκεί και πέρα δεν θα παρέχεται η προστασία. Ποια θα είναι τα όρια αυτού του δικτύου προστασίας. Θα είναι λοιπόν ενδεικτικό ή θα είναι συγκεκριμένο και θα θέτει συγκεκριμένα όρια. Ο πρόεδρος, πριν δώσουμε ξανά το λόγο στην κυρία Λάμπερτ, ε, ορισμένα ερωτήματα απευθύνθηκαν στο Συμβούλιο και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπούργος, εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά την ερώτηση που γίνεται σε μένα. Τα τα άτομα τα οποία προστατεύονται από αυτήν την οδηγία δεν αλλάζουν με την ε, αναδιατύπωσή της. Για τους πρόσφυγες υπάρχει η Σύμβαση της Γενέβης, υπάρχει η Διεθνής Σύμβαση και Αποχρέωση εκ μέρους των κρατών και δεύτερον υπάρχουν οι δικαιούχοι ε, της προστασίας βάση του άρθρου 15 για τους οποίους δεν υπήρχε διεθνής υποχρέωση αλλά είπαμε ότι βάση του κοινοτικού δικαίου έχουν δικαιώματα προστασίας. Πρόκειται για τα άτομα για τα οποία πιστεύουμε ότι αν επιστρέψουν στη χώρα τους, στη χώρα καταγωγής τους, υπάρχει μεγάλος ε, κίνδυνος να πάθουν κάτι σοβαρό κίνδυνος για τη ζωή τους, φερειπίν, να βασανιστούν ή να υποστούν άλλου είδους προβλήματα. Δεν αλλάζουν τα πράγματα με τη νέα πρόταση λοιπόν για αυτούς. Απλώς και μόνο πρέπει να δούμε αν αυτή η δεύτερη κατηγορία προστασίας όσον αφορά τα διάφορα δικαιώματα που παρέχονται είναι τα ίδια. Ούτως ή άλλως, εάν θέλετε κάποιες περαιτέρω εξηγήσει, μπορώ να σας το δώσω και γραπτό συνστήση μεταξύ σα. Η κυρία Γκάν, εκ μέρου τη Επιτροπής. Ευχαριστώ. Είναι αρκετά απλή η ιδέα και είμαστε στη διάθεση τη εισηγήτρια και των σχεδόν εισηγητών για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε κάποιε διατάξει. Η ιδέα όμω δεν είναι να προστατεύσουμε τους πάντες, αλλά να την χορηγήσουμε την προστασία αυτή πλήρως και σε όλους με τον ίδιο τρόπο στην Ευρώπη, σε αυτούς που την αξίζουν και πολλοί την αξίζουν και να την αρνηθούμε σε αυτούς οι οποίοι δεν ε, ικανοποιούν τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν στην οδηγία αυτή και με τρόπο πιο ίσο, αν θέλετε, μεταξύ όλων των μελών που καλύπτονται από αυτή την οδηγία. Ευχαριστώ. Η κυρία Λάμπερτ για την ε, τελική παρατηρήση πριν να ολοκληρωθεί το όλο θέμα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε απολύτω σαφεί. Στην πρόταση αναδιατύπωση, συγγνώμη, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και να ασχοληθούμε είναι αυτά που αποτελούν αντικείμενο τροπολογίας. Εδώ καλύπτονται τα κυριότερα θέματα τα οποία μας απασχολούν, ποιοι είναι δικαιούχοι όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσει, ποιοι όχι και πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς γι' αυτό. Κατά την άποψή μου, εξετάζοντας το άρθρο 15 για σοβαρή βλάβη ή ζημία, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα τροπολόγησής του. Νομίζω ότι σωστά λέγονται αυτά που λέγονται εδώ και ακόμη και αν θέλουμε να το αλλάξουμε το θέμα δεν αλλάζει. Τώρα όσον αφορά τις εθνικές παραδόσεις, τα πλαίσια του άρθρου 4 και με την τροπολογία ε, και στο, στο 3.14 επίσης τα πράγματα σωστά εκφράζονται. Όσον αφορά για το ποιοι είναι οι δικαιούχοι, για ποιους μιλάμε, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η συντριπτική ε, ψηφία που φεύγει από τη χώρα του διοκόμενος πηγαίνει σε μια γειτονική χώρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συνήθως συμβαίνει σε όλους. Φερρυπίν, στο Μπαγκλαντές πηγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από την ε, Μπούρμα. Ε, δεν έχουν φτάσει ακόμα στην Ευρωπαϊκή και θέλουν να καταλήξουν. Θα πρέπει να δούμε επίσης ποια είναι τα κίνητρα του καθενός για να διαλέξει μια χώρα. Οικογενειακοί δεσμοί ή οποιοδήποτε άλλα ε, θέματα ή πρώτα απ' όλα αυτά κυρίως στους διώκονται και μετά να έχουν κοινωνική προστασία και μετά να βρουν εργασία. Επίσης, το θέμα των ασφαλών χωρών. Αυτό δεν έχει μεγάλη σχέση με το θέμα που εξετάζουμε εμείς τώρα. Τώρα, το θέμα του κόστους που ξέρω ότι κάποια έθεσαν. Θα ήταν χρήσιμο, όπως είπε και η Κομισιό, να δούμε την μελέτη επιπτώσεων. Και βεβαίως, προσπαθούμε εμείς μέσω διαφόρων διατάξεων να διευκολύνουμε την πρόσβαση κάποιων ατόμων στην αγορά εργασίας παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορα θέματα θετικά. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε απόλυτα σαφείς. Τι ακριβώς θέλουμε στα πλαίσια της αναδιατύπωσης. Ποιες είναι οι αλλαγές που θέλουμε να εισαγάγουμε. Τώρα, νομίζω ότι μπορεί κάποια μέρη να βελτιωθεί η πρόταση και μετά την συνάντηση που θα έχουμε με τους σκιαδησίτες θα δούμε πώς μπορούμε να τα μελετήσουμε και θα επανέλθουμε. Επίσης, όπως σας είπα, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την συνεκτικότητα της εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Και αυτός είναι ο στόχος κάποιων τροπολογιών που έχουν καταθεί. Τώρα, το θέμα της, ε, ε, του χρονοδιαγράμματος μας ε, ε δόθηκε, είπε καταρχάς κάποιος Ιούνιο, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και θα δούμε οι συντονιστές πώς μπορούμε να συντονιστούμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Λάμπερ. Σχέδιο έκθεσης. 23-24 Ιουνίου, όπως είπατε, αν η συγγήτρια δεν έχει να κάνει κάποια άλλη πρόταση. Και τώρα προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Σημείο 6 ε, και το 6 και το 7 έχουν σχέση μεταξύ τους, διότι ασχολούνται με το σχέδιο σύστασης ε, μετά από δεύτερη ανάγνωση. Έχουμε το σημείο έξω για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το άσυλο. Και πάλι η συγγήτρια είναι η κυρία Τζιν Λάμπερτ και ασχολούμε θα δούμε ένα θέμα κλειδί του προγράμματος της Χάγης. Στις 7 Μαΐου του 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νομοθετικό ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με τροπολογία στην πρόταση Επιτροπής για την δημιουργία μιας υπηρεσίας που θα υποστηρίζει τα κράτη-μέλη για θέματα που αφορούν το κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Έχουμε τώρα την ε, σχέδιο έκθεσης συγγνώμη, το σχέδιο σύσταση κυρία Λάμπερ. για δεύτερη ανάγνωση. Γι' αυτό δίνω αμέσω το λόγο πάλι στην κυρία Λάμπερτ. This is the last issue Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι το τελευταίο θέμα που, για το οποίο θα έχω το λόγο σε αυτή τη συνεδρία Υπομονή, λοιπόν. για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. Πρόκειται για μια υπηρεσία που προτείνεται να δημιουργηθεί με στόχο να φέρει μια πιο δημόσια διάσταση πέρα από τη συνεργασία που ήδη γίνεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη δηλαδή, αλλά να δοθεί και έτσι ψηλότερο προφίλ και πιο συστηματική προσέγγιση βασικά. Στόχος είναι να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ε, ότι η εφαρμογή των διατάξεων περιασύλου να είναι πιο συνεκτική σε όλα τα κρατημέλη. Θα συνεργαστεί δηλαδή με τα κρατημέλη ώστε να βελτιωθεί η εφαρμογή του κεκτημένου περιασύλου. Όσον αφορά τη διαδικασία, Έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά με τους Σκιώδης και με το Συμβούλιο μετά από την πρώτη ανάγνωση. Υπήρχαν διάφορα θέματα, όπως το θυμάστε, γιατί συζητήσαμε τα αποτελέσματα εκείνων των διαπραγματεύσεων στην Επιτροπή. Και διάφορα πράγματα που ήθελε το Κοινοβούλιο όσον αφορά τη λογοδοσία του της υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχέσεις με τον Διευθυντή, για το πώς θα μπορούσε να υπάρχει ένας δεσμευτικός μηχανισμός αλληλεγγύης ανάμεσα στα κρατημέλη. Δεν το καταφέραμε αυτό, αλλά τουλάχιστον κάναμε κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέματα σε σχέση με την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Εκεί συμφωνήσαμε πως θα δημιουργηθεί ένα συμβουλευτικό φόρουμ με εντολή την οποία θα συμφωνήσουμε σε συνεργασία με τον ε, διευθυντή της υπηρεσίας αυτής και άλλα θέματα όπως η σχέση με τρίτες χώρες και ούτω καθεξής. Άποψή μας στο τέλος αυτών των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο ήταν ότι μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτά στα οποία καταλήξαμε. Είχαμε μια ενδεικτική ψηφοφορία, όπως θα θυμάστε, ίσως στις 12 Νοεμβρίου εδώ στην Επιτροπή και μετά στείλαμε μια επιστολή στο Συμβούλιο και τους είπαμε ότι θα πρέπει να επανέλθετε με επιβεβαίωση αυτού του κειμένου και τότε θα ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε και να το συμφωνήσουμε. Η γλωσσολόγοι νομικοί των δύο θεσμικών οργάνων εργάστηκαν επί του κειμένου και οι θέσει του Συμβουλίου εστάλησαν στο Κοινοβούλιο και ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα μόλις, δηλαδή στις 10 Μαρτίου. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε σήμερα μπροστά μας είναι μια σύσταση να προχωρήσουμε και να το εγκρίνουμε, αλλά βέβαια δεν θα είναι σε αυτήν την συνεδρίαση. Θα θέλατε να ελέγξετε ότι το κείμενο του Συμβουλίου, αφού πέρασε και από τους ε, ε, ειδικού είναι το κείμενο το οποίο συμφωνήσαμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και στη συνέχεια να το ψηφίσουμε στην συνεδρίαση της 7ης Απριλίου ώστε να επικυρώσουμε. Ελπίζω πως θα το επικυρώσετε κι εσείς δηλαδή το κείμενο. Φυσικά το Κοινοβούλιο πάντα λαμβάνει τις ε, αποφάσεις του ανεξάρτητα, αλλά αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Σε ευχαριστώ. Η Προεδρία, ο κύριος Μπούργος θέλει να παρέμβει. Ναι, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Για το Συμβούλιο, αυτή η υπηρεσία είναι σημαντική για την ε, βελτίωση της πρακτικής συνεργασίας μέσα στο πλαίσιο της οικοδόμησης ε, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Στο θέμα αυτό, η θέση της Ισπανικής Προεδρίας επί της ουσίας δεν έχει αλλάξει. Δεν έχουμε παρέμβει. Και όπως το είπε και η συγγήτρια, η δουλειά μας και καθήκον μας ήταν να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συμφωνία όσο γίνεται πιο σύντομα, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η υπηρεσία όσο γίνεται πιο σύντομα. Γι' αυτό και ήθελα να ζητήσω από τους ευρωβουλευτές να εργαστούν ε, επιδιώκοντας τον ίδιο στόχο. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή. Μάλιστα. Υποστηρίζουμε τα όσα είπε η Ισπανική Προεδρία, ευχαριστώντας Κνέου για την ε, ταχύρυθμη και αποτελεσματική εργασία της Τζιν Λάμπερ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου. Να σας θυμίσω ότι η Κομισιόν διαβίβασε την περασμένη εβδομάδα μια επίσημη ανακοίνωση, την οποία, ότι δηλαδή υποστηρίζουμε το κείμενο που υιοθετήθηκε μετά από τις εργασίες των νομικών γλωσσολόγων, το κείμενο δηλαδή το οποίο υιοθέτησε το Συμβούλιο στα τέλη του Φεβρουαρίου. Φεβρουαρίου. Merci. Yes, Mr. Buzutil, if you make it short. Ο, Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα ήθελα να συγχαρώ την Jean Lambert για την εργασία της, την θαυμάσια εργασία της την οποία κατάφερε να, να βγάλει, να συγκεράσει από το πακέτο του ασύλου. Συγχαρητήρια λοιπόν για, αυτό το επίτευγμα. Έχω μια παρατήρηση. Στα προηγούμενα σημεία της ημερήσιας διάταξης συζητήσαμε τα δικαιώματα που πρέπει να παράσχουμε στους ετούντες άσυλο, αλλά δεν έχουμε ακόμα συζητήσει το βάρος το οποίο έχουν αναλάβει στις πλάτες τους πολλά κράτη-μέλη, ιδίω της Νότιας Ευρώπης, με την εισρωή των ατόμων αυτών. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια υποκρισία. Από τη μία πλευρά θέλουμε να εδραιώσουμε και να προσφέρουμε περισσότερα δικαιώματα. Από την άλλη πλευρά όμως όταν ζητούμε την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών έτσι ώστε να μοιραστεί το βάρος όλων των εισερχομένων δεν βρίσκουμε ανταπόκριση. Πιστεύω ότι η υπηρεσία αυτή υποστήριξη για το άσυλο θα μπορέσει να επιβάλλει μια δίκαιη κατανομή του βάρους Ε, δεδομένου ότι δημιουργούνται πάρα πολλές ε, δυσκολίες και υποχρεώσεις. Τώρα, δεν έχουμε διευκρινίσει ορισμένα διοικητικά θέματα. Παραδείγματο χάρη, πώ θα επιλεγεί ο διευθυντή, ε, ποιοι θα είναι υποψήφοι, τέτοια διοικητικέ λεπτομέρειε λοιπόν για την υπηρεσία. Το ερώτημα αφορά την Κομισιόν, η κυρία Γκάν. Μα η Κομισιόν περιμένει με ανυπομονησία την υιοθέτηση της πρότασης για να προσχωρήσουμε σε όλες αυτές τις διαδικαστικές ε, εφαρμογές. Γιατί χωρίς νομική βάση δεν μπορούμε να φτιάξουμε την υπηρεσία. Βεβαίως έχουμε ήδη ξεκινήσει μέσω της δημοσίευσης ε, της ε, θέσης του Διευθυντή και περιμένουμε υποψηφιότητες για τον Απρίλιο. Και όταν θα έχουμε την νομική βάση με τα μέλη που θα έχουν ορίσει τα κράτη-μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα προχωρήσουμε στις πρώτες φάσεις για να ε, στελεχωθεί το, η υπηρεσία η οποία θα πρέπει να είναι λειτουργική εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύω του κανονισμού. Γι' αυτό και το περιμένουμε να ξεκινήσει η διαδικασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σχόλια. Ο κύριος Ταβάρες. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος για να πω στην Τζιν Λάμπερτ ότι σύμφωνα με την ενδεικτική μας πληροφορία θα επικυρώσουμε το αρχικό κείμενο και να πω ότι από πλευράς μου πιστεύω πως θα πρέπει να το κάνουμε όσο γίνεται πιο σύντομα, γιατί είναι πολύ καλά προετοιμασμένη αυτή, αυτός ο κανονισμός. Υπήρξε εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στην εισηγήτρια και τους Σκιώδης και το Κοινοβούλιο ήδη έκανε τη δουλειά του ε, και με το παραπάνω για να προχωρήσουμε με ταχύρυθμη διαδικασία, όπως μας ζήτησε και η Σουηδική Προεδρία. Η δικιά μας δουλειά λοιπόν από πλευράς του Κοινοβουλίου έχει γίνει. Το ίδιο ελπίζω να κάνουν και τα άλλα θεσμικά όργανα. Ήθελα μόνο να σχολιάσω αυτό το καλό νέο σε σχέση με την ε, ταχύρυθμη διαδικασία υποψηφιωτήτων για τον ορισμό του διευθυντή της υπηρεσίας αυτής για να πω ότι ζητήσαμε κατά τη διάρκεια του τριμερού διαλόγου, τριμερούς διαλόγου ότι το Κοινοβούλιο θα θελήσει να συμμετέχει στον διορισμό του Διευθυντή. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή κάθε δυνατότητα που μας δίνεται από τα όσα περιλαμβάνονται στην έκθεση της Jean Lambert και θα θέλαμε ε, το πρόσωπο που θα είναι ο διευθυντής αυτού, αυτής της υπηρεσίας να πούμε ότι θα είναι καθοριστική σημασία για τη λειτουργία του, για τη φύση του επίσης και θα θέλαμε αυτός ο άνθρωπος να έρθει εδώ, ο υποψήφιος, και να λογοδοτεί ώστε η κοινωνία των πολιτών να μπορέσει να διαπιστώσει ποιος θα είναι ο χαρακτήρας και η λειτουργία αυτού του θεσμού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις. Θα θέλατε τώρα να κάνετε τα τελικά σχόλια, κύριε Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία να κόψουμε την κορδέλα των εγγενείων της υπηρεσίας αυτής και να δούμε πόσο θα μπορέσει να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη σε αυτό το πολύ σημαντικό τομέα. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, από την Κομισιόν, θα πρέπει και εμείς να βιαστούμε, να προχωρήσουμε στις διαδικασίες μας για την επιλογή του διευθυντή και όλες τις συναφείς ε, διοικητικές λεπτομέρειες. Είχαμε και πρόσφατα τις συζητήσεις για τις σχέσεις του Ευρωκοινοβουλίου με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Άρα λοιπόν θα ήθελα τα μέλη μας να συζητήσουν το θέμα αυτό στις πολιτικές τους ομάδες γιατί θα πρέπει να προχωρήσουμε τώρα στα διαδικαστικά πιστεύω στην αρχή Απριλίου να μπορέσουμε να ψηφίσουμε ε, αυτήν την ε, πρόταση για να προχωρήσουν τα πράγματα γρήγορα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σημειώσαμε το... την τελευταία σας παρατήρηση για τον Απρίλιο και την ακρόαση που πρέπει να κάνουμε, ε, που πρέπει να κάνει η Διευθύνουσα Επιτροπή για τους ε, διευθυντές, την επιλογή διευθυντών. Λοιπόν, προθεσμία υποβολής τροπολογιών 23 Μαρτίου μεσημέρι, 12 η ώρα, ψηφοφορία στην Επιτροπή Λίμπε τον Απρίλιο, 7 και 8 Απριλίου, 7 και 8 Απριλίου, υιοθέτηση στην Ολομέλεια στην, ε, τον Απρίλιο, Απρίλιο. 7-8 Απριλίου στην Επιτροπή και συνεχεία στην Ολομέλεια ολοκληρώσαμε και αυτό. Προχωράμε στο θέμα 7, το οποίο ε, συνδέεται με το θέμα 6, Ευρωπαϊκό Ταμείο της Πρόσφυγης την περίοδο 2008-2013. Η συγητής είναι ο κύριο Κλοντ Μωράε. Δεν είναι παρόν, αλλά τον εκπροσωπεί η κυρία Γκυγιόμ Θέλουμε εδώ να εξετάσουμε ε, σχέδιο ε, πρότασης για δεύτερη ανάγνωση. Σχέδιο σύσταση, συγγνώμη, για δεύτερη ανάγνωση. Η κυρία Γκυγιόμ είναι εδώ και θα μιλήσει εκ μέρου του εισηγητή. Θα προσπαθήσω να τον αντικαταστήσει, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται λοιπόν για μία έκθεση πάρα πολύ σύντομη για θέματα, ε, ασχολείται με θέματα προϋπολογισμού και συνοδεύει την έκθεση της κυρίας Λάμπερ. Περιμένοντας λοιπόν εδώ μία ειδική γραμμή στον προπολογισμό, οι διάφορες, ε, ε, οικονομικές, τα, οι διάφορες οικονομικές ε, δαπάνες θα αναλυφθούν από το Ευρωπαϊκό για τους πρόσχεσεις. Πρόκειται για μια σύντομη πρόταση την οποία κάνει ο και μου ζητάνε να την υποστηρίξετε. Σας ευχαριστώ. Ας ακούσουμε την Προεδρία και την Κομισιό. Έχει κάνει σχόλιο, δεν έχετε σχόλια. Όχι σχόλιο, κανένα σχόλιο, κανένα σχόλιο. Κυρία Παπα-Νικολάου, έχετε το λόγο. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είναι απλό το ζήτημα. Ε, προκειμένου να λειτουργήσει η υπηρεσία η καινούρια πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους πρόσφυγες. Μια προσθήκη μόνο σε σχέση και με μια συζήτηση που είχαμε με συναδέλφους από το δικό μα από τη δική μας πολιτική ομάδα, ε, τίθεται το ζήτημα πώς πάει η χρηματοδότηση από αυτό το ταμείο και αν τα χρήματα αυτά είναι αρκετά και για την νέα αυτή υπηρεσία αλλά και για το πρόγραμμα επανεκατάστασης. Υπενθυμίζω ότι μέχρι πρόσφατα ε, δεν είχαν ε, αξιοποιηθεί όλα τα χρήματα που είχαμε στη διάθεσή μας από αυτό το ταμείο. Πρέπει να έχουμε την προσοχή μας όλοι στραμμένη στα θέματα αυτά φέτος, προκειμένου στο, στο νέο προϋπολογισμό να τα λάβουμε υπόψη μας και να δούμε αν πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Σας ευχαριστώ. Thank you. Any more comments? Άλλα σχόλια παρακαλώ. Όχι, ωραία. Οπότε μπορούμε να ορίσουμε την προθεσμία τροπολογιών 23 Μαρτίου μεσημέρι, 12 η ώρα, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Απρίλιο 7 και 8 και υιοθέτηση στην Ολομέλεια του Απριλίου. Πολύ ωραία. Moving to point number Προχωρούμε λοιπόν στο σημείο 8. Προχωρούμε τώρα. Προχωρούμε. στην εδραίωση στο, ε, ε, πρόγραμμα της ε, επανεγκατάστασης θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης. Έχουμε τροπολογίες και συμβιβαστικές τροπολογίες τις οποίες ε, πρέπει να εξετάσουμε και την προθεσμία υποβολής τροπολογιών που προτείνεται να είναι... Α, λέει 2 Μαρτίου λέει ο πρόεδρος. Ναι. Α, πέρασε. Και τώρα συζητούμε το σημείο 8 και το σημείο 9 για την επαναγκατάσταση. Η συγητής είναι ο κύριος Ταβάρες και μετά θα δώσω το λόγο στην Προεδρία και στο Συμβούλιο. Εισηγητή, παρακαλώ, κύριε Σταβάρε. Σε κατάσταση συζητούμε. Σας ευχαριστώ. Νομίζω πως θα πρέπει από κοινού να εξετάσουμε αυτά τα σημεία. Θα θυμάστε τις ε, συζητήσεις που είχαμε και την ε, κοινή συζήτηση που είχαμε πρόσφατα για αυτές τις δύο εκθέσεις, θα πρέπει να λάβουμε απόφαση γιατί υπάρχουν κάποιες τροπολογίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων που αποζημιώνει τα κράτη για τις δαπάνες τις οποίες ε, προκλήθηκαν ε, μέσα στη διάρκεια επανεγκατάστασης των προσφύγων σε τρίτες χώρες και Ταυτόχρονα πιστεύουμε πως μια γραμμή του προπολογισμού και μια αποζημίωση προς τα κάτι μέλη δεν αρκεί για να έχουμε μια διαδικασία επαγκατέσταση των προσφύγων που να είναι στεναρή και φιλόδοξη και ότι θα ήταν ε, πολύ σημαντικό και κατά τη, όπως φάνηκε και κατά τη διάρκεια της ε, Σουηδικής Προεδρίας πρόκειται για περίπου 5.000 πρόσφυγες που εγκαθίσατε τη ίωσες στην Ένωση. Πιστεύουμε πω αυτό δεν αρκεί ωστόσο. Θα θέλαμε να υπάρξει μια έκθεση πρωτοβουλία και το Κοινοβούλιο να συγκεντρώσει τις ιδέες του και να ε, χαράξει μια πορεία ώστε να έχουμε ένα καλό κοινό πρόγραμμα επανακατάστασης των προσφύγων. Είναι λοιπόν μια έκθεση πρωτοβουλία ε, σε συνεργασία με του σκιώδει εισηγητές ήταν εξαιρετική και επικοδομητική. Είχα πολλές ευκαιρίες για να ακούσω τις ιδέες των συναδέλφων. Λάβαμε διάφορες τροπολογίες, εννέα για τη συναμπόφαση και 140 τροπολογίες για την ε, έκθεση πρωτοβουλίας οι περισσότερες από αυτές είτε δεν υπήρχε πρόβλημα είτε μετά από μια συνεδρίαση με τους κοιόδης εισηγητές θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε συμβιβαστικές προτάσεις που θα ικανοποιούν τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Για να σας δώσω κάποια παραδείγματα, ένα από τα πράγματα που ζητούσαμε ήταν να ε, την επιλογή των ε, κατηγοριών να γίνονται μέσω μιας πρώτης αξιολόγησης ε, που θα γίνεται από την ΑΚΝΟΥΡ και έπειτα ε, να έχουμε και διάφορες ε, περιφερειακές κατηγορίες στις οποίες θα δίνει προτεραιότητα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, για ορισμένες δηλαδή περιοχές του πλανήτη. Αυτά κάνα τα εξετάσαμε σε μια πρώτη συζήτηση και θεωρήσαμε πως θα πρέπει να είναι επαρκή και τα κονδύλια γιατί το θέμα της επανεγκατάστασης των προσφύγων πολλές φορές έχει να κάνει με θέματα ανθρωπιστικά και θα πρέπει να προσέξουμε τους ανθρώπους που δεν εντάσσονται σε αυτές τις ε, περιφέρειες, ε, σε αυτές τις κατηγορίες, μπορεί να είναι στην Αφρική ή στην Μέση Ανατολή, σε οποιαδήποτε περιφέρεια του πλανήτου όπου εμείς ε, ορίζουμε τις αιτήσεις τις προτεραιότητές μας αλλά μπορεί να προέρχονται από διάφορες καταστάσεις και θα πρέπει αυτό να αναγνωρίζεται από την Υπατερμοστία. Αρμοστία. Ε, ορίζονται οι ευαίσθητες ε, κατηγορίες ανθρώπων όπως τα παιδιά, οι γυναίκες, οι αυτοί που χρειάζονται βοήθεια, οι ασθενείς, οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε στρατόπεδα προσφύγων και που δέχονται ένοπλες επιθέσεις ή εκεί όπου έχουν υπάρξει φυσικές καταστροφές και ας πούμε, στρατόπεδα προσφύγων όπου έχει γίνει, έχουν γίνει πλημμύρες ή άλλου είδους φυσικές καταστροφές, όπου δεν μπορούν δηλαδή να παραμένουν εκεί ή σε κάποιες ε, περιπτώσεις δεν μπορούμε καν να προβλέψουμε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και άλλες ε, κατηγορίες. Αυτές ήταν οι πιο σημαντικές ε, συζητήσεις που έγιναν εδώ. Υπάρχουν και άλλες ιδέες ανακατηγορία, <coughs> αλλά σήμερα έχουμε φτάσει σε μία συνένεση όσον αφορά τους ανθρώπους που θα έπρεπε να έχουν την προτεραιότητα στην επανεγκατάσταση. Αυτοί οι οποίοι έχουν επιβιώσει από βία ή βασανιστήρια, ε, ευάλωτες κατηγορίες ανθρώπων, άνθρωποι που χρειάζονται επιγόντως επανεγκατάσταση λόγω ανάγκης προστασίας, άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχθεί απειλές ε, στη σωματική τους, για τη σωματική τους ακεραιότητα, ή ανθρώπους οι οποίοι ε, είναι υπό απειλή ένοπλης επίθεσης ή άλλες ανθρωπιστικές καταστάσεις που δεν έχουν εδώ προβλεφθεί αλλά μπορεί να εμπίπτουν στις ε, προτάσεις των κρατών μελών για την κατάσταση ανθρώπων που βρίσκονται σε πήγουσα ανάγκη. Έπειτα, το θέμα της διαφοροποίησης, δηλαδή θέλουμε με βάση μια ανάγκη η οποία εκφράστηκε από την ίδια την Κομισιόν, από τον ε, επίτροπο τον τότε επίτροπο μας είχε πει λοιπόν πως χρειαζόταν να γίνουν περισσότερο ώστε να ε, ενταχθούν τα κράτη-μέλη σε αυτό το πρόγραμμα και ο τρόπος στον οποίο σκεφτήκαμε για να γνωστοποιήσουμε το πρόγραμμα αυτό στα κράτη-μέλη ήταν να δώσουμε αυξημένες ε, αποζημιώσεις τα πρώτα δύο χρόνια γιατί κάθε φορά είναι αυτό πιο δαπανηρό τα δύο πρώτα χρόνια για τα κράτη-μέλη δηλαδή να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα επανεγκατάστασης σε προσφύγων. Γιατί θα πρέπει να προσληφθούν ε, άνθρωποι, να στελεχωθούν υπηρεσίες ή ακόμα και πολλές φορές να κατασκευαστούν και υποδομές. Καταλήξαμε λοιπόν ότι θα πρέπει σαφώς να πούμε ότι αυτό το μέτρο θα πρέπει να εφαρμόζεται και να υιοθετηθεί από τα κράτη-μέλη στην κατασκευή οικοδόμηση ενός βιώσιμου προγράμματος επαναγκατάστασης, ώστε δηλαδή για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τα κράτη-μέλη είναι σημαντικό να τους γνωστοποιήσουμε πως είναι ανάγκη να κάνουν ε, αυτό που άλλα κράτη-μέλη που έχουν παράδοση στην επαναγκατάσταση των προσφύγων και που σίγουρα έχουν πληρώσει τις ηθικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά τη βοήθεια προς τους πρόσφυγες, κάνοντας προγράμματα ορισμένα από τα οποία είναι εξαιρετικά και μας έχουν εμπνεύσει όσον αφορά αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας. Είναι ανάγκη λοιπόν και αυτά τα κράτη-μέλη να έχουν ε, κάποια κονδύλια στη διάθεσή τους για την ε, ε, υλοποίηση ενός βιώσιμου προγράμματος για κατάσταση προσφύγων. Εδώ νομίζω πως εύκολα θα βρούμε συμβαστικέ λύσει ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη και στην έκθεση πρωτοβουλία. τα πράγματα προχωρούν καλά. Εδώ προσπαθούμε να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών, τους Δήμους, ε, αλλά και διάφορες ενώσεις που μπορούν να συμμετέχουν στην προσπάθεια επανεγκατάστασης και έχουμε μεγάλη συνένεση. Αυτό αποδεικνύεται και από το ότι σχεδόν δεν υπήρξαν τροπολογίες. Ε, να έχουμε δηλαδή μια μόνιμη ομάδα επανεγκατάστασης με το κατάλληλο προσωπικό που θα μπορεί να προβαίνει σε όλη αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στην υπατερμοστία, τα κράτη-μέλη, την κοινωνία των πολιτών και άλλες ε, οργανισμούς που ασχολούνται με τους ε, πρόσφυγες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν πέρα από το κονδύλι του προπολογισμού να υπάρχουν οι απαραίτητοι μόνιμοι ανθρώπινοι πόροι ε, που θα ασχολούνται με το θέμα αυτό. Υπάρχει επίσης και νομίζω πως ήδη έχουμε κάνει διάκριση από την επανεγκατάσταση, την επανατοποθέτηση των προσφύγων, η επανεγκατάσταση των προσφύγων που έρχονται από τρίτες χώρες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ε, πτυχές που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Είναι δηλαδή κάτι, εντάξει το λέω κάπως απλουστευτικά, αλλά εμπίπτει και στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής. Το Κοινοβούλιο θέλει δηλαδή να συμμετέχει στον καθορισμό των προτεραιοτήτων και προσφέραμε το Κοινοβούλιο στην να γίνει κοινή ε, συνεδρίαση μεταξύ των Επιτροπών ΛΥΜΠΕ, Ανάπτυξης και Εξωτερικών να δούμε δηλαδή ποιος ε, θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολόκληρο τον κόσμο θα πρέπει να έχουμε μια γενική πρακτική για τους πρόσφυγες εντός των εσωτερικών συνόρων της Ένωσης. Και πιστεύω πως όλες οι διακυβερνητικές οργανώσεις, η ΜΚΟ και η η Κομισιόν εργάζονται με αυτούς τους όρους και γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι ακριβώς σημαίνει επανεγκατάσταση, επανατοποθέτηση ακόμα και αν ε, αναγνωρίζουμε ότι είναι το ίδιο σημαντικές και οι δύο αυτές πτυχές. Τώρα, έχουμε και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των ε, μέτρων. Ήδη υπήρξε ένα άνοιγμα στην τελευταία συζήτηση όσον αφορά τις ε, εξουσιοδοτήσεις. Θα πρέπει να δούμε όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις της ίδιας της Κομισιόν για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Εμείς θεωρούμε πως αυτές εμπίπτουν ε, ε, στις ε, εξοδοτημένες ενέργειες της Κομισιόν. Από πλευράς της Κομισιόν φαίνεται πως ένα κομμάτι αυτών όλων θα πρέπει να γίνει υπό τη συναπόφαση, αλλά θα πρέπει ακριβώς να γίνει ο διαχωρισμός του τι εμπίπτει στη συναπόφαση και τι όχι. Ήδη υπήρχε εδώ καλή συνένεση και ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να εκφράσει τη βούλησή του να προχωρήσει γρήγορα και στεναρά σε αυτή την πολιτική. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας δε στο ότι κατά βάση θα πρέπει να κάνουμε μια awareness day, μια ημερίδα συνειδητοποίηση εδώ στο Κοινοβούλιο στις 15 Απριλίου. Εμείς γνωρίζουμε ακριβώς τι θα πει επανεκατάσταση και επανατοποθέτηση, αλλά θα πρέπει να το γνωρίζουν και όλοι οι βουλευτές του σώματος. Πρόκειται για μέτρα τα οποία θεωρούνται βιώσιμα και ανθρώπινα όσον αφορά τη μεταχείριση των προσφύγων που δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσή τους ούτε στις χώρες διέλευσης μπορούν να παραμείνουν και έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες από την ύπατη τερμοστια Άρα λοιπόν στις 15 Απριλίου, παραλαμβάνω, θα έχουμε αυτή την ημερίδα ενημέρωσης και συνειδητοποίησης με διάφορες ΜΚΟ εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ταβάρες. Ο κύριος Μπούργος, Ισπανική Προεδρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα αναφερθώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για του Πρόσφυγες, δεδομένου ότι είναι το αντικείμενο της συναπόφασης. Πήραμε την πρόταση της Επιτροπής στο Συμβούλιο. Η αξιολόγησή μας είναι σχετικά θετική, γενικά, η αξιολόγηση των κρατών μελών, διότι κατανοούμε ότι επειδή υπάρχει ήδη η δυνατότητα χρηματοδότησης κάποιων κρατών για την επανεγκατάσταση, το να προχωρήσουμε σε συντονισμό και να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σημαίνει ότι προφανώς υπάρχει για το θέμα αυτό τη θέμενη αξία. Άρα η αξιολόγησή μας είναι θετική. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να μελετήσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σημειώσαμε ότι βασικά και εσείς κινείστε στην ίδια γραμμή με αυτές τις τροπολογίες και θα διευκολυνθεί η δουλειά μας έτσι, μελετώντας τις. Είχαμε κάποιες ανεπίσημες επαφές με τον εισηγητή και πιστεύουμε ότι στα πλαίσια των ε, προθεσμιών θα μπορέσουμε να σας εκφράσουμε την πλειοψηφική άποψη του συμβολίου σε σχέση με τις ε, τροπολογίες όσον αφορά τα πάγια ετήσια ποσά ή τα οικονομικά κίνητρα για τις χώρες που θέτουν σε εκκίνηση τη διαδικασία επανεγκατάστασης. Τώρα, όσον αφορά τις τροπολογίες διαδικασίας, θα τις μελετήσουμε με μεγάλη προσοχή. Και πιστεύω ότι σύντομα Επίσης και για αυτές θα μπορέσουμε να έχουμε τη θέση της πλειοψηφίας των κρατών μελών και να τη συζητήσουμε με τον εισηγητή. Προς το παρόν αυτό που μπορώ να σας πω είναι η προτεραιότητά μας. Η διαδικασία να είναι πρακτική και αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η Κομισιό, η κυρία Μαρτίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την υποστήριξή του στην πολιτική της επανεγκατάστασης. Αυτή η προσέγγιση του προκύπτει από το σχέδιο έκθεσης. Επίσης ευχαριστώ και τα άλλα μέλη του σώματος ε, για τις τροπολογίες τους. Θα ήθελα να σχολιάσω λίγο τις ε, τροπολογίες που αφορούν τις αποφάσεις για αυτό το Ταμείο Προσφύγων. Καταρχάς, στόχος της πρότασης της Κομισιόν. Ποιος ήταν ο στόχος. Καταρχάς έχουμε μία απόφαση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων που επιτρέπει την οικονομική ενίσχυση για την κατάσταση. Επιτρέπει λοιπόν ε, την οικονομική στήριξη ε, ευάλωτων ομάδων, γυναικών, παιδιών που έρχονται ε, από άλλες χώρες υπό το πλαίσιο της επανεγκατάστασης. Ορισμένοι τώρα ενδιαφερόμενοι μας είχαν πει ορισμένοι φορείς ότι αυτά τα κριτήρια δεν έχουν αρκετή ευελιξία και μας ζήτησαν να υιοθετήσουμε μια νέα προσέγγιση και να αυξήσουμε την ευελιξία αυτής της πολιτικής επανεγκατάστασης και να κάνουμε μία πιο γενική συζήτηση για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της επανεγκατάστασης. Γι' αυτό ακριβώς εμείς προτείνουμε στην πρότασή μας μία ευέλικτη προσέγγιση η οποία δεν υπησέρχεται τόσο πολύ σε λεπτομέρειες ανακατηγορία αλλά αφήνει ανοχτό το ενδεχόμενο μιας δημόσιας συζήτησης με την κοινωνία των πολιτών, με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί όχι, για να καθορίσουμε τα στατηγικά κριτήρια. Το σχέδιο γνωμοδότησης ε, λοιπόν ε, του εισηγητή και ακόμα περισσότερο οι τροπολογίες οι οποίες αυξάνουν τα κριτήρια στον κατάλογο ενδέχεται να αλλάξουν τελείως ε, την ε, ουσιαστική προσέγγιση και να δημιουργήσουν εκτενείς ε, καταλόγους ή κριτήρια τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν κάθε κατηγορία και υποκατηγορία ατόμου που εμπίπτει στην επανεγκατάσταση. Γι' αυτό σας παρακαλώ να σκεφτείτε με πολύ προσοχή την ορολογία και τους ορισμούς που έχουν ήδη υιοθετηθεί για τα άτομα που εμπίπτουν στο καθεστώς επανεγκατάστασης. δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ μεγάλο κατάλογο κατηγοριών, διότι έτσι περιορίζουμε ακόμα περισσότερο την ευελιξία μας. Και τότε όλη αυτή η συζήτηση δεν έχει και νόημα. Εκτός όμως από αυτόν τον μεγάλο κατάλογο προτείνεται και αλλαγή διαδικασιών. Για με, εγώ δεν καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο να καταλάβω γιατί θέλουμε να καθιερώσουμε διαδικασίες οι οποίες δεν μας επιτρέπουν κανένα περιθώριο υιοθέτηση νομικών πράξεων. Αυτό το οποίο θα αποφασίζεται ε, κάθε χρόνο είναι προφανές. Με το Κοινοβούλιο, με το Συμβούλιο λοιπόν εξετάζουμε τις τροπολογίες. Ε, δεν λέω, αλλά πιστεύω ότι η ουσία των τροπολογιών αλλάζει τελείως την αρχική προσέγγιση. Επίσης προτείνει τον ορισμό μιας συγκεκριμένης νομικής πράξεως για να καλυφθεί αυτό το θέμα. Dedicated Act, λοιπόν, Procedure, μια διαδικασία συγκεκριμένης νομικής πράξης και πιστεύω ότι αυτό θα περιορίσει πάρα πολύ την ευελιξία μας. Εμείς θέλουμε, δεδομένου ότι μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους πρόσφυγες, να διατηρήσουμε την ευελιξία αυτού του τομέα, αυτής της πολιτικής. Δεν καλύπτει μόνο την επανεγκατάσταση, αλλά και πολλά άλλα θέματα προσφύγων δεν θέλουμε με κανέναν τρόπο η πολιτική της επανεγκατάστασης να υπονομεύσει, να διακυβεύσει τις εξαιρετικές πολιτικές που έχουν ήδη καθιερωθεί σε άλλα θέματα προσφύγων. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις, δεν λέω, αλλά πάντοτε πρέπει να έχουμε κατά νου το βασικό μας στόχο στο θέμα της οικονομικής ενίσχυσης ε, που, που μπορεί να δοθεί σε κράτη-μέλη τα οποία επιλέγουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επανεγκατάστασης. Ήδη έχουμε εδώ δεχθεί ευέλικτα, ευέλικτες διατάξεις, ευέλικτα μέτρα για τα κράτη-μέλη αυτά. Η μόνη ανησυχία που έχουμε είναι ότι πρέπει να καθιερώσουμε ξεκάθαρα κριτήρια έτσι ώστε τα κράτη-μέλη που θέλουν να συμμετάσχουν και να δεχθούν οικονομική ενίσχυση να ξέρουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Σαφή κριτήρια λοιπόν. Ακριβής ορολογία, ακριβής νομική βάση, γιατί εδώ πρόκειται για λεφτά, τα οποία θα ξοδέψουμε, για να μην μπλέξουμε με το ελεγκτικό συνέδριο. Όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις που έκανε ο εισηγητής σε αυτό το πεδίο, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής θα αποφασίσει ε, την ατζέντα, το πρόγραμμα και πιστεύουμε ότι έτσι θα διευκολυνθεί όλη η διαδικασία επαναγκατάστασης η οποία θα γίνει και πιο σαφής. Το Ευρωκοινοβούλιο βεβαίως συμμετέχει στις συζητήσεις και έχουμε μια ανοιχτή προσέγγιση στη συζητήση μας με το σώμα. Ε, όλοι είμαστε ενδιαφερόμενοι, μας αφορά όλους αυτό το θέμα. Ένα άλλο σημείο το οποίο δεν αναφέρθηκε αλλά υπάρχει στην έκθεσή μας είναι η οικονομική ενίσχυση. Χρησιμοποιούμε εδώ ένα ταμείο το οποίο χρησιμοποιείται και για άλλες δραστηριότητε. Δηλαδή, αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο δεν ασχολείται μόνο ή δεν καλύπτει μόνο, δεν χρηματοδοτεί μόνο την επανεγκατάσταση, αλλά και πολλές άλλες δραστηριότητε. Γι' αυτό στις ε, μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει να καθιερώσουμε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο, μία γραμμή συγκεκριμένη που να καλύπτει αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Εμείς ε, δεν μπορούμε να ε, ε, επηρεάσουμε ή να διαμορφώσουμε τις δημοσιονομικές προοπτικές αλλά πιστεύω ότι μια συγκεκριμένη γραμμή ε, το στον προπολογισμό στα πλαίσια της δημοσιονομικής προοπτικής θα μας διευκολύνει στην καλύτερη λειτουργία του Ταμείου. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητής, αλλά σας παρακαλώ να είσαστε σύντομοι για να σεβαστούμε και το χρονοδιάγραμμά μας. Έχουμε ακόμα τους συντονιστές για μισή ώρα, τουλάχιστον. Αντώνιο Μασίπ, παρακαλώ. Πολύ σύντομα, συμφωνώ με αυτά που λέτε, Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι συμφωνώ απόλυτα και υποστηρίζω απόλυτα τον εισηγητή στο θέμα αυτό. Όχι μόνο για τα θέματα τα οποία μελετάμε και τροποποιούμε, αλλά και για το πνεύμα εργασίας. Δηλαδή, διότι Έχουμε πάρα πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των σκιωδών και του εισηγητού. Θα ήθελα επίσης να τον ευχαριστήσω για την ε, φαντασία που επιδεικνύει για να μας δώσει παραδείγματα, για να μας πει πώς έχουν τα πράγματα και αλλού. Στην Ασία, στη ΣΥΠΑ, στην Καναδία καταβάλει λοιπόν μία προσπάθεια η οποία πιστεύω ότι είναι μία, ένα πολύ αξιόλογο προηγούμενο για τις εργασίες που αναλαμβάνουμε στο Κοινοβούλιο. Σήμερα, όλο το απόγευμα, είδαμε ότι μπορούν να υπάρχουν ε, ε, διαφορές ε, σημασιολογικές, ορολογίας, νομικής φύσης μεταξύ των μελών της Επιτροπής μας, αλλά κάθε φορά βλέπουμε όλο και λιγότερες ιδεολογικές διαφορές. Και είδαμε ότι πραγματικά όλοι βασικά σεβόμαστε στην ε, Ευρώπη με κοινέ αρχές τους πρόσφυγες, αυτούς τους οποίους πρέπει να προστατεύσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κατορθώσαμε τελευταία χρόνια και δεν ήταν ένα πνεύμα που ίσχυε εδώ και χρόνια στο Κοινοβούλιο. Προσπαθούμε λοιπόν με προσέγγιση μεταξύ όλων ημών στις πολιτικές ομάδες να κάνουμε την μετανάστευση μία μετανάστευση νόμιμη και κυρίως για θέματα πολιτικής μετανάστευσης, μιλάω για την οικονομική. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει, λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη το Συμβούλιο, να εργαστεί και με μεγαλύτερη ταχύτητα, για να μην χαθεί η σημασία του ότι κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν προσεγγίζοντας οι μεν τους δε και τις ιδεολογίες του Κοινοβουλίου με αυτές του Συμβουλίου να προχωρήσουμε γρήγορα. Δεν μπορεί για τόσο σημαντικά θέματα να ε, καθυστερεί πάρα πολύ η κάθε Προεδρία. Ευχαριστώ. Κύριος Παπα-Νικολάου. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς να συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή. Πράγματι με τον κύριο Ταβάρες έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και θέλω να τον ευχαριστήσω γι' αυτό. Κατατέθηκαν και από την δική μας πολιτική ομάδα ε, μια σειρά τροπολογιών. Οι περισσότερε από αυτές στόχο έχουν να ενισχύσουν το κείμενο, πάντα σε συνεργασία με τον εισηγητή. Ε, θέλω να δώσω έμφαση σε ορισμένα σημεία ε, σύντομα. Το πρώτο είναι ότι πράγματι με αυτήν την έκθεση και την ιδέα πρωτοβουλία και την απόφαση που πρέπει να λάβουμε ε, στόχο έχουμε να πείσουμε περισσότερα κράτη-μέλη να εμπλακούν στη διαδικασία. Σωστά πρέπει να ε, δίνουμε έμφαση σε θέματα ανθρωπιστικά. Σωστά πρέπει να δώσουμε έμφαση και στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Και σε όλα αυτά δεδομένο είναι ότι και αλληλεγγύη θέλουμε να υπάρξει μεταξύ των κρατών μελών και ε, όσο γίνεται να αναπτυχθεί αυτή η πρωτοβουλία. Στη συζήτηση που είχαμε όλο αυτό το διάστημα και γι' αυτό ε, κάνω την πρώτη μου παρατήρηση αναφέρομαι στην τροπολογία 17 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο των Προσφύγων για την απόφαση πρέπει να λάβουμε και στις τροπολογίες 2 και 37 στην έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας προχωρήσαμε σε μία ε, τροπολογία η οποία αναφέρεται σε μια πολύ απλή σκέψη η οποία όμως αποτελεί μεγάλη ανάγκη. Πράγματι έχουμε ανάγκη για επανεγκατάσταση γιατί όμως αυτή η επανεγκατάσταση δεν πρέπει να ισχύει και να ανοίξουμε αυτό το πρόγραμμα που έχουμε και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου υπάρχουν ε, πράγματι πολλοί πρόσφυγες με τεράστιες ανάγκες που και αυτοί έχουν ανάγκη να λύσουν τα προβλήματα για την διαβίωσή τους και την ομαλή ένταξή τους στις κοινωνίες των κρατών μελών. Και στο σημείο αυτό ε, αποδέχομαι αυτό που λέει και η Επιτροπή για το διαφορετικό ε, ορισμό, το resettlement δηλαδή και το reallocation. Στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο όμως για τη μετανάστευση και το άσυλο, ο ορισμός είναι ενιαίος. Και εν πάση περιπτώσει, με εξαίρεση στο πιλωτικό πρόγραμμα στη Μάλτα που είχαμε μέχρι σήμερα, πρωτοβουλίες της Επιτροπής για θέματα τέτοια, για ε, ε, επαναπροώθηση δηλαδή προσφύγων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε διοργανωμένα και εδώ ενισχύω και εγώ την τοποθέτηση του κυρίου Μπουζουτήλ προηγουμένως σε σχέση με την υποκρισία που κάποιες φορές δείχνουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ακριβώς λοιπόν για αυτούς τους λόγους και πάντα θέλοντας να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια και σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα ε, στις εκθέσεις αυτές και στην προσπάθεια πράγματι την πολύ σοβαρή που γίνεται, αυτό που εμείς ε, τοποθετούμε είναι ακριβώς η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε συνολικά το θέμα, να έχουμε δίκαιη κατανομή των βαρών σε όλα τα κράτη-μέλη συνολικά για το θέμα των προσφύγων και βεβαίως η περιβόητη αλληλεγγύη στην οποία συνεχώς αναφερόμαστε. Ω εκ τούτου, θέλω να παρακαλέσω όλου του συναδέλφου να αντιληφθούν αυτή την ανάγκη, ιδίω για τι χώρε εκείνες οι οποίε επιβαρύνονται κατά τρόπο δυσανάλογο και κατά τρόπο με τον οποίο δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν από μόνες τους, αναφέρομαι ιδίως στον Ευρωπαϊκό Νότο, προκειμένου να αξιοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων για να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο τα ζητήματα της ελληνικής και της συμπαράστασης μεταξύ των κρατών μελών. Περιμένω τις τοποθετήσεις και του Συμβουλίου και της Επιτροπής και βεβαίως των συναδέλφων ε, και βεβαίως είμαστε ανοιχτοί σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο, αν για κάποιο λόγο ε, επειδή είχαμε μια τέτοια ε, συζήτηση προηγουμένως με τους, στη συνάντηση που είχαμε τον εισηγητή και τους υπόλοιπου συναδέλφους που είναι οι αν υπάρχει κάποιο θέμα που στο νομικό σκέλος πρέπει να δούμε, ευχαρίστως να το αντιμετωπίσουμε. Το βασικό όμως είναι να αντιληφθούμε σε πολιτικό επίπεδο ότι πρέπει επιτέλου να δούμε συνολικά το θέμα. βεβαίω να έχουμε συμπαράσταση για ανθρωπιστικά θέματα. Βεβαίω όμω αυτό να το κάνουμε όχι μόνο για τι τρίτε χώρε, να το κάνουμε και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση για τι χώρε που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Ένα δεύτερο, μια δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να πω και αλλάζω θέμα για να κλείσω. Ε, και, στην, και η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. αλλά και ε, σε συζητήσεις που είχαμε και με τις ΗΠΑ με μια πολύ ωραία ε, έτσι, τηλεδιάσκεψη που οργάνωσε ο εισηγητής και τον ευχαριστούμε, ε, τονίζεται κάθε φορά και η ανάγκη συμπαράσταση στα θέματα αυτά και από φορείς οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι φορείς, είναι ιδιωτικοί φορείς και δεν αναφέρομαι βεβαίως σε εταιρείε, αναφέρομαι σε ιδρύματα, αναφέρομαι σε οργανισμούς, οι οποίοι, σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις, σε οργανισμούς οι οποίοι πολλές φορές για πολλούς λόγους ανθρωπιστικούς εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες. Γι' αυτό έχουμε καταθέσει στην έκθεση πρωτοβουλίας ε, ιδίας πρωτοβουλίας μία τροπολογία για τη συνδρομή του ιδιωτικού τομέα. Αν η φρασιολογία προκειμένου να έχει τη συνένεση όλων πρέπει να εμπλουτιστεί κατά κάποιο τρόπο, ευχαρίστως να το κάνουμε προκειμένου και πάλι όλοι όσοι θέλουν να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια να είναι ελεύθεροι να το κάνουν και εμείς να τους ανοίγουμε ακόμη περισσότερο το δρόμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Um, ως σχέδιο συγκέντρια για τις Πάσης θέλει και εγώ για την εξαιρετική του έκθεση και την δουλειά που έκανα συγχαρώ τον εισηγητή. Υποστηρίζουμε πλήρως την έκθεσή του. Απλώς θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις για τρία σημαντικά σημεία. Πρώτα απ' όλα, διαφάνεια των κριτηρίων. Εδώ μιλάμε για ομάδες Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ διφωνείς για το πώς θεσπίζονται τα κριτήρια που αφορούν αυτές τις ομάδες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συμμετέχει σε όλη τη διαδικασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα έσπιση των κριτηρίων και μην το αφήνουμε μόνο στους άλλους. Δεύτερον, Τώρα, η εποπτεία του πώς αντιμετωπίζουν το θέμα της επανεγκατάστασης οι χώρες υποδοχής και πώς λειτουργεί όλη η διαδικασία καθώς και η διαδικασία ενσωμάτωσης των ατόμων που επεγκαθίστανται είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελέγχουμε για να μπορούμε να δίδουμε συμβουλές για πώς μπορούν να βελτιώσουν κάποια πράγματα τα κράτη-μέλη. Είναι επίσης σημαντικό όλο το σύστημα να λειτουργεί σωστά. Τρίτη παρατήρηση. Καλούμε επιγόντως τα κράτη-μέλη να θεωρήσουν την ναι, κατάσταση των ατόμων τα οποία ζητούν ε, να επανεγκατασταθούν και ξέρουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι απλή. Πώς το Συμβούλιο θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη για να επιτύχουν αυτά τα προγράμματα τα άτομα τα οποία ζητούν να επανεγκατασταθούν, να επανεγκατασταθούν. Ευχαριστώ, κύριος Μπόνς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν συμφωνώ με τον εισηγητή και το σχέδιο έκθεσής του, διότι πάει πολύ μακριά. Ζητά να προσέξουμε όλους σε όλες τις ε, ευάλωτες εμάς του κόσμου. Να μιλήσουμε για το Πακιστάν, τη Σομαλία, το Ιράν, τον Ταρφούρ, το Ιράν, αλλά δεν μπορούμε στην Ευρώπη να δεχθούμε τη μισό κόσμο. Από όλη την οικουμένη. Δεν συμφωνώ λοιπόν με την έκθεσή του. Ζητώ λοιπόν τουλάχιστον κατανότατο όριο, συγγνώμη, με επίγοντα χαρακτήρα να δεχθούμε, δεχόμεθα 2.000 άτομα. Διαφορετικά, αν κάνουμε ό,τι λέει στην εκθεσή του, θα αντιμετωπίσουμε την πλήρη κατάσταση. Uh, Ο κύριος Λαμπρινίδης, μια εκθέση Ένις Πλάσ. Ήταν απολύτω σαφέ ότι ζητήσαμε μηχανισμό επανεγκατάστασης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξαν να το γνωρίσουν αυτό και η Κομισιόν και το Συμβούλιο και έκαναν πρόταση για την εμπακατάσταση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για κάτι το οποίο ως ιδέα είναι απολύτως ευγενής και την υποστηρίζουμε, αλλά αυτό δεν μπορεί να επισκιάσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου του προηγούμενου Μαΐου να ζητήσει με ευρύτατη ε, πλειοψηφία έναν ενδοκινοτικό μηχανισμό για το θέμα αυτό. Αυτό τι σημαίνει. Ότι επειδή φάνουν τώρα με πρόταση η Κομισιόν και το Συμβούλιο ε, για κοινοτικού μηχανισμού δεν θα πρέπει να ανησυχεί το Κοινοβούλιο. Τι θα πρέπει να έχουμε μία πρόταση πρωτοβουλίας διαφορετική μόνο για την ενδοκινοτική επανεγκατάσταση. Η απάντησή μου είναι όχι. Και ο λόγο είναι, η αιτία είναι, ότι αυτή η ειδική πρόταση και αυτό ο ειδικό μηχανισμό σημαίνει ότι θα δοθούν και κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων. Εάν όλα τα κονδύλια ε, του Ταμείου αυτού θα πρέπει να δοθούν για την επανεγκατάσταση των εξοκοινωτικών, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στα άλλα ε, δύο όργανα ότι εμεί ζητήσαμε κάτι και ενδοκινοτικό Και αν πάρω όλα τα λεφτά στην για την πρόταση τη δική του, δεν θα μείνει τίποτα για τη δική μα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην υποχωρήσει για να τα πω τα πράγματα ως έχουν και να μην αφήσουμε το Συμβούλιο και την Κομισιό να κοφεύσει σε αυτά τα που είχαμε προτείνει πέρσι. Θα πρέπει να πούμε ότι επενθυμίζουμε στο Συμβούλιο και στο Επιτροπή ότι θέλουμε να υπάρχει και ενδοκοινοτικός μηχανισμός επανεγκατάστασης και ζητούν τα κονδύλια τα οποία ε, θα δοθούν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων να, να ε, προβλέψουν και αυτό το μηχανισμό τον ενδοκινοτικό και όχι να πάνε μόνο σε αυτά τα οποία υποστηρίζει η Κομισιό και το Συμβούλιο. Όπως λέει και ο εισηγητής, σωστά και ανθρώπινα είναι τα κριτήρια τα οποία θεσπίζονται, αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι και οι πρόσφυγες των δικών μας κοινοτικών χωρών μπορούν όταν είναι δυνατόν και απαραίτητο να επωφεληθούν από τα ίδια κριτήρια. Ευχαριστώ κύριε Μπουσούτιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να συγχαρώ τον Γουι Ταβάρης για την έκθεσή του και να υποστηρίξω την έκθεση του όσον αφορά τη δημιουργία του κοινού προγράμματος επαναγκατάστασης, αλλά θέλω επίσης να υποστηρίξω τον συνάδελφο Παπα-Νικολάου και Λαμπρινίδη, όσον αφορά το εσωτερικό την εσωτερική μοιρασιά του φορτίου εντό τη Ένωση. Δεν ακούσαμε καμία αιτιολόγηση, καμία λογική αιτιολόγηση, Πρόεδρε, γιατί να υπάρχει η δυνατότητα επανεγκατάστασης απέναντι στι τρίτε χώρε, αλλά όχι ανάμεσα στα κράτη-μέλη τη Ένωση. Δεν υπάρχει καμία λογική αιτιολόγηση γι' αυτό μέχρι στιγμή. Μας είπαν ότι υπάρχει διαφορά στη διατύπωση, επανεγκατάσταση είναι για εκτό Ένωση και επανατοποθέτηση για ε, εντό Ένωση. Αλλά αυτά είναι μόνο και μόνο σημασιολογία, λέξεις διαφορετικές. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται όμως για αυτά. Ο κόσμος θέλει αλληλεγγύη πραγματική. Αλλά δυστυχώ, όπω είπε σωστά ο κύριος Λαμπρινίδη, αυτή η έκθεση αγνοεί την εσωτερική αλληλεγγύη παντελώ. Εγώ θα ήθελα να πω το εξή και θα ολοκληρώσω. Πώ μπορούμε εμεί, ιδιαίτερα οι ευρωβουλευτέ από την Ελλάδα, από την Κύπρο, από την Ισπανία, από την Ιταλία, από τη Μάλτα, τη χώρα μου, να πάμε στου ε, ψηφοφόρου μα και να του πούμε: Κοιτάξτε, αν δείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλι έφτιαξε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάσταση, αλλά όχι για μα, είναι για τι τρίτε χώρε μόνο. Μα είναι γελίο αυτό. Δεν είναι δυνατόν να διαβάσουμε εμεί τέτοιο πολιτικό μήνυμα. Και αν και ο Σταύρο έχει απόλυτο δίκιο όσον αφορά τα οικονομικά του ζητήματο, εγώ να προσθέσω ότι και οι πολιτικέ πτυχέ είναι ακόμα πιο σημαντικέ. Δεν είναι μόνο δηλαδή ε, θέμα χρημάτων. Θα πρέπει να δώσουμε ένα πολιτικό μήνυμα στι χώρε μα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται όχι μόνο για την επανεκατάσταση εκτό Ένωση, αλλά και εντό Ένωση. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ η κυρία Χίρς. Σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ ως σκιώδης εισηγήτρια. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη θαυμάσια και επικοδομητική συνεργασία. Ειδικά σε αυτό το θέμα πρέπει να διευκρινίσουμε τις διαφορές ε, εάν υπάρχει επανεγκατάσταση ατόμων ε, όπως θα πρέπει να υπερισχύσει μία αλληλεγγύη ή εάν υπάρχει ε, μία επανατοποθέτηση του ατόμου αυτού σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη περιοχή Ας μην ξεχνάμε, relocation και, ενδοκινοτική Ναι, και ενδοκινοτική μετεγκατάσταση. No. Ναι. Resettlement και relocation, ε, ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες γυναικών και παιδιών. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα τα άτομα αυτά να εισέλθουν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους υποστηρίξουμε με το πλαίσιο που έχουμε τη δυνατότητα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μπερδέψουμε την ενδοκινοτική μετεγκατάσταση με την εγκατάσταση από τρίτες χώρες ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε όλο αυτό το πρόγραμμα του resettlement, της επανεγκατάστασης, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και την υποδομή των σχολείων, την υποδοχή των υπηρεσιών υγείας και για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια μακροπρόθεσμη προστασία στα άτομα αυτά που την δικαιούνται. Γι' αυτό υποστηρίζω ολόθερμα την ε, ε, έκθεση του κυρίου Ταβάρης. Κύριε Παπαδοπούλου, σύντομα παρακαλώ. Και τον κύριο Λαμπρινίδη. Όταν μιλούμε για πρόσφυγες δεν δικαιόμαστε ως Ευρωπαίοι βουλευτές να έχουμε επιλεκτικές ευαισθησίες. Πρέπει να υπάρχει δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων και οπωσδήποτε κοινοτική αλληλεγγύη και προς τους ε, ανθρώπους που προέρχονται από τρίτες χώρες, αλλά κυρίως και προς τον Ευρωπαϊκό Νότο. Α μην ξεχνάμε ότι οι πρόσφυγε υπάρχουν σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Οι Ευρωπαίοι πολίτε δεν έχουν μόνο δικαιώματα, ε, μόνο υποχρεώσει έχουν και δικαιώματα και θα συμφωνήσω απόλυτα με την άποψη που έχει πει ο κ. Λαμπρινίδη ότι επιβάλλεται να υπάρχει ένα ενδοκοινωτικός μηχανισμό επανεγκατάστασης και εντό της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η κοινοτική αλληλεγγύη πρέπει να υπάρχει και σε οικονομικών επίπεδων και σε επίπεδο πολιτική, αλλά και σε επίπεδο πολιτικών που να αφορά του πρόσφυγε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ένις Πλάσου. Και εγώ πολύ σύντομα. Κατανοώ το σκεπτικό και πιστεύω ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία. Οι διαφορές όμως ποικίλουν και οι δυσκολίες ποικίλουν μεταξύ του resettlement και του relocation ενδοκινοτικά και από τρίτες χώρες. Εγώ πρότεινα ένα συμβιβαστικό κείμενο που είναι ένα πολύ απλό εκτιμώντας για να κάνουμε μία σαφή αναφορά στην ουσία και Εάν λοιπόν εσεί θέλετε να σταματήσουμε τη συζήτηση πολύ γρήγορα, αλλά η πρόταση που έχω κάνει εγώ για ένα επιπλέον εκτιμώντας είναι σαφέστατη και σύντομη. Ο κύριος Μπούργος από το Συμβούλιο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Πάλι ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που κάνατε για μας παρατήρησα και σημείωσα όλες τις θέσεις, θα τις συζητήσω με τους συναδέλφους όπως πρέπει. Έγινε συγκεκριμένη ερώτηση, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη για να συμμετάσχουν σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επαγγελματάστασης. Η αλλαγή αυτού του Ταμείου για πρόσφυγες θα χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο κατά κύριο λόγο, διότι προβλέπεται χρηματοδότηση και υπάρχει και η δυνατότητα συμμετοχής στον σχεδιασμό αυτού του ευρωπαϊκού προγράμματος. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι οι συζητήσεις που έγινε σε πολιτικό επίπεδο στο Συμβούλιο, όχι τόσο για την πρόταση αυτή συγκεκριμένα, αλλά γενικά για την εγκατάσταση ότι η ιδέα που επικράτησε είναι ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν ε, βάσει βούλησης του κράτους μέλους. Σε αυτό συμφωνεί η πλειοψηφία. Και αυτό θα ισχύει και για την έκθεση αυτή και για οποιοδήποτε πρόταση υποβληθεί στο μέλλον. Εμείς κατανοούμε ότι η πρόταση της Κομισιό αναφέρεται στην επανεγκατάσταση από άτομα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό την περίπτωση μελετήσαμε. Τώρα, αν υπάρχει τροπολογία προς άλλη κατεύθυνση, όπως είναι η υποχρέωσή μας, θα τη μελετήσουμε. Αλλά μέχρι τώρα αυτό το οποίο κάναμε ήταν να μελετήσουμε την πρόταση που είχαμε μπροστά μας. Επίσης, θα ήθελα να πω παράλληλα αυτά, ότι στο παρόν ταμείο για τους πρόσφυγες υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης για περιπτώσεις της εσωτερικής μετεγκατάστασης, αν θέλετε. Οποιαδήποτε κράτο μέλο λοιπόν μπορεί να υποφεληθεί αυτή τη δυνατότητα που παρέχεται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μαρτίνη, παρακαλώ σύντομα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη, διότι υπενθύμησε η Προεδρία ότι είναι εθελούσιο αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και τι σημαίνει ότι θα δοθεί περισσότερη χρηματοδότηση για κάποιες κατηγορίες ατόμων που θέλουν να επεγκατασταθούν. Αυτή είναι η κατάσταση που ισχύει σήμερα. Δεν αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα, το ταμείο. Είναι κάτι το οποίο προσβλέπεται στο Ταμείο Προσφύγων. Αυτό το οποίο προβλέπουμε να κάνουμε είναι να θεσπίσουμε τις κατηγορίες με διαφορετικό μηχανισμό ετησίως κάθε χρόνο. Να μην έχουμε ε, συγκεκριμένες κατηγορίες πάγιες. Και βεβαίως θα δώσουμε χρηματοδότηση χωρίς να θέλουμε να επιβάλλουμε σε κανένα να δεχθεί άτομα. Έχει εθελούσιο χαρακτήρα αυτό το μέτρο. Θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το παρόν Ταμείο Προσφύγων η οικονομική ενισχύριση για ενδοκοινοτική μετεγκατάσταση είναι κάτι το οποίο έχουμε. Δεν έχω μπροστά μου όλα τα άρθρα του δημοσιονομικού κανονισμού. Είναι κάτι το οποίο προβλέπεται στα πλαίσια του Ταμείου Προσφύγων. Μπορούμε να υποστηρίξουμε αν αποφασίσουν να κάνουν ενδοκοινοτική μετεγκατάσταση ατόμων. Τρίτον, πιστεύω ότι είναι σωστό να λέμε ότι η Επιτροπή κόφευσε στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιδείξει αλληλεγγύη. Λήφθησαν διάφορα μέτρα και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την ε, εσωτερική επαναγκατάσταση ατόμων από τη Μάλτα, στο οποίο συμμετέχουν πολλά κράτη-μέλη. Πρόκειται για πιλωτικό πρόγραμμα, προς το παρόν ισχύει για τη Μάλτα πρώτα. Ε, πρόκειται ε, σε θελούσια βάση πάντα για 50 άτομα, αλλά πάντα με την υποστήριξη, όπως λέμε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και αυτή τη στιγμή γίνεται και μελέτη για τις επιπτώσεις του προγράμματος για να δούμε εάν μπορούμε να προβλέψουμε ένα μηχανισμό ε, καταμερισμού του βάρους και η Επιτροπή πάντα έλεγε ότι αυτό ενδεχομένως θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω στου πιο φιλόδοξε τέτοιου είδου πρωτοβουλίε. Θέλω να επιθυμίσω όμω ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα και δεν είναι αληθέ ότι η Επιτροπή δεν κάνει τίποτα για την, ε, στα πλαίσια της ενδοκινοτικής ελεγγύης. Αλλά αυτή τη στιγμή συζητούμε εδώ το θέμα της ε, επανεγκατάστασης και αλλάζουμε αν θέλετε τους κανόνες για να υποστηρίξουμε τις τρίτες χώρες. Πράγμα το οποίο ενδεχομένως θα έχει και σημαντικές επιπτώσεις ε, για τις ε, ε, χώρες οι οποίες πρέπει να επιμεριστούν το βάρος και μπορούν να βοηθηθούν κατά κάποιο τρόπο οι χώρες υποδοχής στην, ε, κοινοτική, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνάδελφος ασχολείται με αυτό το θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι τώρα θέλει να προσθέσει τίποτε. Όχι. Αυτό. Ο κύριος Σταβάρες. Συγγνώμη. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Λαμπρινίδη. Ο κύριος Σταβάρες. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Παρά το γεγονό ότι είναι δύσκολο αυτό, γιατί τέθηκαν πολλά θέματα. Πιστεύω. Τέλο αν θα μιλήσω πορτογαλικά γιατί πρέπει να συγκεντρωθώ. Και στη μητρική μου γλώσσα τα λέω ε, καλύτερα, αλλά ίσως κάποια στιγμή κάνω και κάποια παρατήρηση στα αγγλικά. Λοιπόν, για να απαντήσω πρώτα απ' όλα σε κάποια θέματα τα οποία ανέφερε και η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Είναι αληθές ότι οι δύο διαφορετικές αυτές κατηγορίες, οι μόνιμες, δηλαδή ανθρωπιστικού χαρακτήρα για άτομα τα οποία ήταν θύματα βίας, βασανιστήριων, ε, σεξουαλικής ε, συμπεριφοράς κάποιων και οι αιτήσιες κατηγορίες αν θέλετε που είναι θέμα στρατηγικής της κοινότητας για το που θέλουν να παρέμβουν δεν είναι ταυτόσιμες. Και όπως είπε η κυρία Μαρτίνη υπάρχουν κάποιες που έχουν ε, την ε, το προτέρημα να είναι μόνιμες για ηθικούς και ανθρωπιστικούς λόγους ως κατηγορίες και τις άλλες είναι θέματα στρατηγική τα οποία μπορεί να σκεφτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για δύο-τρία χρόνια. Δεν το κάνουμε εμεί μόνο αποκλειστικά. Ο Καναδά, Φερρυπίν, αποφασίζει για τρία-τέσσερα-πέντε χρόνια ότι θα επικεντρωθεί στην Κεντρική Αμερική ή στην ακτή του Ελεφαντόβοντο ή σε κάποια περιοχή τη ε, Ασία που θέλει, που έχουν ε, κάποια ανάγκη. Σε πέντε χρόνια μπορεί να αποφαρίσει ότι στρατηγικά του συμφέροντα είναι να αλλάξει. Συγχρόνως όμως έχει και κατηγορίες που δεν χρειάζεται να είναι ρητά οι κατηγορίες που έχουν εγγραφεί στην ορολογία της ΥΠΑ αρμοστίας. Μπορεί ο καθένας να έχει κατηγορίες στην ε, δική του νομοθεσία που να συμπεριλαμβάνουν ε, ε, άμεση μνήα των πρεσβειών και τι μπορούν να κάνουν σε διάφορες χώρες του κόσμου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο προτείνουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε συνδυασμό της πολιτικής στρατηγικής που θέλουμε να ακολουθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα επανέλθουμε. Και αυτό, αν θέλετε, είναι από τη φύση του κάτι το οποίο άπτεται και της εξωτερικής πολιτικής μας. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και την ΑΦΕΤ και την ΔΕΒΕ ως επιτροπές. Τώρα, υπάρχουν και οι ανθρωπιστικές μας δεσμεύσεις και πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτές. Το γνωρίζουμε όλοι. Προφανώς, εδώ έχουμε ένα θέμα χρηματοδότησης αυτής της προσπάθειας θέλουμε να ολοκληρώσουμε. Και ξέρουμε όλοι ότι το 2013 είναι το κρίσιμο έτος. Όταν, ε, ολοκληρω... Όταν ε, τελειώσει το 2013 θα χρειαστούμε πάλι ένα νέο ταμείο για τους πρόσφυγες. Τώρα, αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι λιγότερα κονδύλια, αλλά λιγότεροι πρόσφυγες. Αυτή τη στιγμή 20 εκατομμύρια ετησίως δαπανώνται και πρέπει να πω ότι οι ανάγκες μπορεί να είναι πολύ περισσότερες. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας και αυτό είναι κάτι το οποίο κατά την διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας το είπε το Συμβούλιο ότι θέλουμε να προσφέρουμε κατάσταση σε 100.000 πρόσφυγες ετησίως. Και τώρα εποφελούμε για να απαντήσω σε κάτι που ο κύριος Μπρόνς, αλλά δεν είναι εδώ. Εδώ δεν μιλούμε για ευάλωτα άτομα ανά τον κόσμο, αλλά για άτομα ευάλωτα που βρίσκονται σε διάφορα ε, ε, σε καταστάσεις σύμφωνα με, που έχουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε καταγράψει με την βοήθεια της ΥΠΑΣ της αρμοστίας. Και εάν θέλει να ανταποκριθεί στα αιτήματα και στι ανάγκε τέτοιων ατόμων μπορούμε να το κάνει στα ευρωπαϊκά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλούμε λοιπόν για κάτι το οποίο είναι ρεαλιστικό και για κατηγορίε ατόμων που έχουν οριστεί με πολύ περιοριστικό και συγκεκριμένο τρόπο. Και εδώ θα προσπαθήσω να απαντήσω στο θέμα της ενδοκινοτικής σε σχέση με την εξοκινοτική επανεγκατάσταση. Όταν άρχισα εγώ να δουλεύω αυτή την έκθεση, πήρα τους ορισμούς έτσι όπως υπήρχαν. Το resettlement έτσι όπως το ορίζει η ύπατη αρμοστία, τα έγγραφα της Κομισιό, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι άτομα τρίτων χωρών που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι άτομα, ε, και, εδώ, και για αυτά τα άτομα είχαμε τη νομική βάση. Δεν είχαμε να κάνουμε με άτομα ε, των οποίων ενδοκινοτικών αν θέλετε για την επανεγκατάστασή τους. Εμείς ε, για αυτό το θέμα μπορούμε να έχουμε μία πάρα πολύ καλή πολιτική ευρωπαϊκή για πρόσφυγες και για άτομα που ζητούν προστασία. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι τα Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων καλύπτουν τις ανάγκες και των δύο κατηγοριών ατόμων, όπως ελέγχθηκε από την Κομισιό. Τι είναι σημαντικό να κάνουμε εμείς, δεδομένου ότι εμείς εδώ συμφωνούμε ότι είναι σημαντική και η ενδοκινοτική κατάσταση. Τι χρειαζόμαστε θα πρέπει να έχουμε και για αυτό το θέμα σαφή πολιτική βούληση. Οι πολιτικές οι οποίες προβλέπονται για την κατάσταση εξοκοινωτικών ατόμων είναι καλές και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και για θέματα με την κατάσταση ενδοκοινωτικά κάποια από τα μέσα για τον ε, κοινοτικό έλεγχο είναι σωστά. Απλώς θα πρέπει εμείς να εκφράσουμε την πολιτική μας βούληση ότι δεν πρόκειται για θέμα ε, μετάθεσης του βάρους, αλλά είναι θέμα ε, καταμερισμού του βάρους. Όταν κάποιος ε, έρχεται στην κοινότητα, δεν λέει από πριν θέλω να πάω ειδικά στην Ελλάδα ή ειδικά στη Μάλτα. Λέει θέλω να πάω στην κοινότητα, στην, Ευρωπα... στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συμφωνώ με αυτά που είπαν και ο κύριος Παπα-Νικολάου και ο κύριος Λεμπρινής και ο κύριος Μπουσούτιλ, καθώς και η κυρία Παπαδοπούλου. Αλλά πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω και κάποιους περιορισμούς εδώ. Και ίσως θέσουμε εν κινδύνο το resettlement χωρίς να κατορθώσουμε να τίποτα για το relocation. Εάν μπορέσουμε να βρούμε πώς θα μπορέσουμε από κοινού να χρησιμοποιήσουμε τις δύο αυτές έννοιες, νομίζω ότι ό,τι κάνουμε για, τις για την εξοκοινοτική μετανάστευση μπορούμε να το εφαρμόζουμε για την ενδοκοινοτική. Και πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε μια συνενετική λύση. Δηλαδή, στο, στην έκθεση για το resettlement να πούμε ότι μας ενδιαφέρει και το relocation. και η πολιτική reallocation δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι εντελώς αντίθετο από την ε, εξοκοινοτική ε, με την κατάσταση. Εγώ μπορώ να δεχθώ λοιπόν την πρόταση που έκανε η Ζανίν. Λοιπόν, ξαναγυρίζω στα πορτογαλικά. Η κυρία Μαρτίνη, και τελειώνω με αυτήν την παρατήρηση, ερωτά τελικά το εξής. Εάν Έχουμε κατάλογο μονίμων κατηγοριών, τι κατορθώνουμε. Ακούστε, δεν μπορούμε να έχουμε σαν shopping list μία μόνιμη κατηγορία και ο καθένας ε, ε, για τους πρόσφυγες να λέει από αυτή την ε, κατηγορία ποιον διαλέγει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ευέλικτος ο κατάλογος αυτός. Αυτό δεν σημαίνει ε, ούτως ή άλλως ότι η κατη, οι κατηγορίες αυτές, οι λίστες αυτές είναι δεσμευτικέ. Είπαμε ότι όλα γίνονται βάσει της εθελούσια πολιτικής του κάθε κράτου. Και βεβαίω, κάθε χρόνο έχουμε τον κατάλογο, κάθε χρόνο υπάρχουν ορισμοί, βλέπουμε ποιοι είναι οι πρόσφυγες και από πού προέρχονται και βεβαίως όπως έχουμε συμφωνήσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι άπτεται και του καταλόγου των ε, προσφύγων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτως ή άλλως πρέπει να συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία και έχουμε την σχετική ψηφοφορία, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε τι είδου συγκεκριμένα μέτρα προβλέπει η Κομισιόν για να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική resettlement, για να δούμε Ποια από αυτά μπορούμε να τα βάλουμε από κοινού σε όλη τη διαδικασία της συναπόφασης και ποια όχι. Πιστεύω λοιπόν ότι με αυτές τις απαντήσεις απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους. Ε, που έλαβαν το λόγο για να συζητηθεί το θέμα αυτό. Κύριε Λαμπρινίδη, μην ξαναρχίσουμε τη συζήτηση, λέει ο Πρόεδρος. Πολύ σύντομα, για να απαντήσω στην Κομισιό. Είπατε ότι δεν κοφεύσατε στις, ε, στα αιτήματά μας. Δύο πράγματα ζητήσαμε. Υποχρεωτική αλληλεγγύη. Δεύτερον, για ενδοκινοτική επανεγκατάσταση. Άρα λοιπόν, ποιες δύο προτάσεις μας ε, εισακούστηκαν. Καμία από τις δύο. Κοφεύσατε και στις δύο. Όπως και το παράδειγμα της Μάλτας, η εθελούσια ε, αλληλεγγύη ισοδυναμεί με τίποτα, διότι οι χώρες δεν θέλουν να, την παράσχουν. Και τέλος κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με την ανάλυση σας μεν, αλλά επανέρχομαι στο οικονομικό μου αίτημα και θέλω αυτή η τροπολογία να συμπεριληφθεί. Είπατε ότι 100.000 πρόσφυγες ε, θα έπρεπε να είχαν τύχη αυτή της επανεγκατάστασης και ζητάτε σε τρία χρόνια 50.000, 15.000 ε, ευρώ σε αυτό το τριετές διάστημα για κάθε πρόσφυγα. Ε, το, το, προσπάθησα να υπολογίσω τον, ε, το κόστος στο κινητό μου ε, υπολογιστή αλλά δεν, δεν μπορούσα να χωρέσει τον αριθμό. Είναι τόσο μεγάλος 100.000 επί 15.000. Εάν λοιπόν δεχτούμε τις προτάσεις ως έχουν τότε τα κονδύλια που θα διατηθούν θα είναι μηδενικά. Μηδέν για την επανεγκατάσταση, ε, για το θέμα αυτό για το οποίο υποτίθεται και έγινε η Κομισιόν. Λοιπόν, δεν μπορεί να περάσει μια τέτοια πρόταση. Ε, παρόλο, φοβόσαστε την άποψη του Συμβουλίου και δεν είναι δυνατό να περάσει μια τέτοια πρόταση η οποία θίγει ολόκληρο το Ευρωκοινοβούλιο. να απαντήσω στο οικονομικό, στο οικονομική, στην οικονομική παρατήρηση. Βεβαίως 100.000 πρόσφυγες ανά χρόνο δεν είναι αριθμό τον οποίο φίβρα εγώ, τον είπε η Σουηδική Προεδρία. Εάν επανεγκαταστήσουμε 100.000, δεν πρόκειται περί αυτού, 4.500 περίπου το χρόνο καλύπτει αυτή η επανεγκατάσταση. Άρα λοιπόν τα, τα πραγματικά στοιχεία μας αφορούν. Εάν επιτύχουμε να διπλασιάσουμε τον αριθμό αυτό από 4.500 ας πούμε σε 9, πιστεύω θα έχουμε επιτύχει. Οπότε χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο ταμείο να υποστηρίξει αυτή την στρατηγική Τώρα, εάν από τις 5.000 πάμε σε 100.000 ε, πρόσφυγες, θα χρεοκοπήσουμε παταγωδός. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το θέμα είναι ε, να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ε, επανεγκαθιστάμενους σε μας μέσα στην κοινότητα, όχι παγκοσμίω. Άρα λοιπόν δεν είναι τέτοια τεράστια διάσταση του θέματος. Η επανεγκατάσταση όπως ε, έθιξε η κυρία Μαρτίνες, έχει θετική επίπτωση ε, μακροχρόνια, μακροπρόθεσμα, διότι εάν εφαρμόζεις την επανεγκατάσταση εξ αρχής και τους μοιράζεις και αυτό μπορεί να γίνει με συντονισμένο τρόπο. Τους μοιράζεις με ισόρροπο τρόπο ε, στην Ήπειρό μας, μειώνεις την πίεση μακροπρόθεσμα. Βεβαίως, <clears throat> αυτή δεν είναι μια βραχυπρόθεσμη λύση, αλλά μακρυπρόθεσμα πρόθεσμα μπορούμε να βοηθήσουμε την επανεγκατάσταση με δύο τρόπους. Ε, να βελτιώσουμε τις διατάξεις που υπάρχουν και δεύτερον οι πρόσφυγες που έρχονται να επανεγκατασταθούν αμέσως ε, ε, σε ένα αποφασισμένο δίκτυο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ξεπεράσαμε το χρόνο μας. Είχαμε μία περιστατωμένη και εις βάθος συζήτηση και τώρα να, να, δούμε το χρονοδιάγραμμα. Ως προτείνεται, η ψηφοφορία προσανατολισμού θα γίνει τον Απρίλιο 7-8. 7-8 Απριλίου. Η ψηφοφορία επιβεβαίωσης ε, Απρίλιο 27 και 28. Και η οθέτηση του σχεδίου ψηφίσματο θα γίνει στο Στασβούργο το Μάιο. Εντάξει. Ωραία, οπότε είμαστε έτοιμοι για τους συντονιστές. Ζητώ τους ε, συντονιστές να μείνουν στην αίθουσα και όλοι οι άλλοι να φύγουν, παρακαλώ, διότι είναι και κλεισμένο των θυρών. The committee will be resuming its works tomorrow. Και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας ως Επιτροπή αύριο στις 9 με την υπόλοιπη ατζέντα. Okay.